ε, αυτή τη στιγμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Κομισιόν ε, πριν ε, από τις καλοκαιρινές διακοπές για τη δάση παγκοσμίω και για την αποψήλωση των δασών και τι συνέβη οπότε με όλα που έγιναν φέτος το καλοκαίρι είναι πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση με την Επιτροπή μας Έχουμε την κυρία Σαμάκερ από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι διευθύντρια ε, για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη από την DG ε, Περιβάλλοντος, από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Είναι πολύ σημαντική η μάχη κατά της αποψήλωσης. Έχετε 10-15 λεπτά το πολύ για την παρουσίαση της ανακοίνωσης και μετά θα κάνουμε το catch the eye με τα μέλη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ε, ευχαριστώ που μου δείτε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτή την ανακοίνωση. Όπως είπατε είναι πολύ επίκαιρο το θέμα και εκτιμάμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια για τις δικές μας προτάσεις. Τι θα κάνω στα 10 λεπτά που έχουμε. Θα σας παρουσιάσω το τι συμβαίνει, τις ε, κινητήρες δυνάμεις που αφορούν την αποψήλωση, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε και κυρίως τις δράσεις τις οποίες προτείνουμε εμείς να υιοθετηθούν. Uh, uh, Τα δάση είναι κάτι αναγκαίο. Δεν χρειάζεται να το υπογραμμίσουμε στην Επιτροπή σας και βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο. Έχουμε μια διεθνή δασική κρίση θα μπορούσα να πω. Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, είδαμε τις ε, πυρκαγιές ε, στον ε, Αμαζόνιο που έφτασαν στα σέλιδα των εφημερίδων και που ανησυχούν τον κόσμο και μετά είχαμε και τις πυρκαγιές και στο Κονγκό, στην Αφρική, σε ένα σωρό μέρη. Η αποψήλωση των δασών είναι σοβαρή. 1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών περιοχών έχουμε χάσει από το 1990 μέχρι το 2016 είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο μεγάλο είναι αυτή ε, η επιφάνεια. Ο Επίτροπος Βέλα χθε ε, προσπάθησε να το κάνει κατανοητό λέγοντας ότι ο πλανήτης χάνει περίπου το αντίστοιχο 800 ποδοσφαιρικών γηπέδων κάθε ώρα, κάθε μέρα. Τα περισσότερα από όσα συμβαίνουν ε, σε θέματα απώλειες των δασών ε, δεν είναι στην Ευρώπη, είναι εκτός Ευρώπη Στην Ευρώπη έχουμε θετική τάση μεταξύ του 1990 και του 2015. Καταφέραμε να αυξήσουμε τις δασικές μας περιοχές στην Ευρώπη. Ουσιαστικά έχουμε περισσότερα δάση. Σχεδόν έχει αυξηθεί η δασική, έχουν αυξηθεί οι δασικές περιοχές σε εμβαδόν ίσο με την επιφάνεια τη Ελλάδα. το 20% των, ε, το 12% όλων των εκπομπών ε, αερίου του θερμοκηπίου προέρχονται από τη χρήση γης και την αλλαγή χρήση γης λόγω κυρίως ε, της ε, αποψήλωσης των δασών. Ε, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή μετά από τα ορυκτά καύσιμα αερίου του θερμοκηπίου η αποψήλωση και τα δάση που περιέχουν τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο γιατί αυτό έχει σημασία, είναι σαφές το 30% της ε, γης καλύπτεται από δάση. Όπως είπαμε η βιοποικιλότητα είναι σημαντική και τα δάση είναι σημαντικά για την κλιματική αλλαγή αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι και ένα 6 ε, δισεκατομμύρια άνθρωποι, 25% του παγκόσμιου πληθυσμού βασίζεται στις δασικούς, στους δασικούς πόρους ε, για τη ζωή του. Ε, η δασική κρίση λοιπόν συνεπάγεται και η κοινωνική κρίση. Χάνεται ένα δάσο, ο κόσμο χάνει τα προστοζήν και αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο, που πλήττονται περισσότερο, είναι οι πιο φτωχοί, οι αυτόχθονε πληθυσμοί σε πολλέ ε, αναπτυσσόμενε χώρε. Τι προκάλεσε τώρα την κατάσταση, κατά κύριο λόγο, θα λέγαμε ότι η γεωργική επέκταση είναι αυτή που ε, είναι η βασική αιτία της αποψήλωσης των δασών. Το 80% της αποψήλωσης των δασών οφείλεται στην μετατροπή δασών σε γεωργικές γέες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι ε, ο μόνος λόγος. Ε, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η αστική επέκταση, η ανάπτυξη υποδομών και η εξόρυξη μεταλλευμάτων. Και αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και έμεσε αιτίε ε, σε διάφορε χώρε, αδύναμε πολιτικέ, αδύναμη διακυβέρνηση, ε, έλλειψη ε, επενδύσεων, ασαφή γεωκτητικά καθεστώτα και δικαιώματα, παράνομες δραστηριότητες. Απαιτείται λοιπόν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει να παίξει κάποιο ρόλο σημαντικό. Γιατί το λέμε αυτό, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε και κατανάλωσε περίπου το 1 τρίτο των προϊόντων ε, που, του παγκοσμίου εμπορίου που προέρχονται από την αποψήλωση. Ε, φινικέλαιο, κρέας, ε, προϊόντα υλοτομίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και την ευθύνη αλλά και την ευκαιρία να επηρεάσουμε το τι συμβαίνει στην παραγωγή αυτών των αγαθών. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η αποδάσωση είναι ένα πρόβλημα κάποιου άλλου που συμβαίνει κάπου αλλού στον πλανήτη. Είναι δικό μα πρόβλημα. Είμαστε και εμεί κομμάτι του προβλήματο και με αυτή την ανακοίνωση προσπαθούμε να επιτύχουμε να, είμαστε και, να γίνουμε και μέρο τη λύση. Η πρόεδρο τη Κομισιόν, Βαντρελάιαν, είπε ότι θέλουμε να γίνουμε παγκόσμιοι ηγέτε στη βιοπικιλότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ε, ως στόχο να ηγηθούμε ε, του κόσμου στη μάχη κατά της αποψήλωσης των δασών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η νέα ανακοίνωση θα μας βοηθήσει να ξεκινήσουμε. Φυσικά τα δασικά ζητήματα μας αποσχολούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Το 2003 είχαμε ένα σχέδιο δράσης κατά της παράνομη υλοτομίας. Ε, ήταν γνωστό ως FLECT και μετά το 2008 σε μια ανακοίνωση είχαμε θέσει φιλόδοξους στόχους για την καταπολέμηση της αποψήλωσης των δασών. Είχαμε πει ότι θέλουμε να σταματήσουμε την απώλεια των δασών μέχρι το 2030 παγκοσμίω και να μειώσουμε την αποψήλωση των τροπικών δασών κατά 50% ε, ε, έως το 2020. Αυτό είναι ουσιαστικά αύριο και όλοι ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν ε, επιτυχάνουμε αυτά που θέλουμε. Πρέπει να επιταχύνουμε λοιπόν ε, τις δράσεις μας, ε, να αλλάξουμε την προσέγγιση μας και να εμπλουτίσουμε το εργαλειοθήκη μας. Γι' αυτό έχουμε αυτή την ανακοίνωση για να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή δράση, ώστε να σώσουμε τα παγκόσμια δάση. Να έχουμε στα χέρια μας περισσότερα εργαλεία, ώστε να εμποδίσουμε τα σημερινά δάση και τα αυτοφύη δάση να καταστραφούν και να αυξήσουμε την δασοκάλυψη παγκοσμίω. Έχουμε εντοπίσει πέντε προτεραιότητες, προτείνουμε 36 δράσεις ε, σε αυτές τις πέντε προτεραιότητες και το πιο βασικό είναι ότι η ανακοίνωση περιλαμβάνει και ένα παράρτημα με συγκεκριμένες συστάσεις για τις αρχές αλλά και για τους ενδιαφερομένους στην κοινωνία των πολιτών και για τη βιομηχανία. Η λέξη κλειδί που θα ήθελα να συσχετήσω εγώ με αυτή την ανακοίνωση είναι ότι πρέπει να εργαζόμαστε ως εταίροι. Εταιρική σχέση είναι η λέξη κλειδί συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιαφερομένων αλλά και εταιρική σχέση με τους εξωτερικούς ε, συνεργαζόμενους, με τις ε, χώρες παραγωγής και άλλες χώρες κατανάλωσης. Οι πέντε προτεραιότητες ε, που έχουμε εντοπίσει συνοψίζονται με πέντε λέξεις κλειδιά. Θέλουμε να εργαστούμε στην πλευρά της ζήτησης, στην πλευρά της προσφοράς, θέλουμε να ενισχύσουμε την διεθνή συνεργασία, να εξετάσουμε τη χρηματοδότηση για όλα αυτά και την έρευνα και τις επενδύσεις για καλύτερη ενημέρωση στη μάχη κατά της αποψήλωσης των δασών. Τα λίγα λεπτά που μου απομένουν θα τα χρησιμοποιήσω για να δούμε λίγο πιο λεπτομερώς τις δράσεις που προτείνουμε, ξεκινώντας με τη μείωση της κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ευρωπαϊκού αποτυπώματος. Δηλαδή εδώ έχουμε τέσσερις τομείς δράσης που έχουμε εντοπίσει. Πρώτον, η σημερινή Επιτροπή λέει ότι πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να ρυθμίσουμε ε, με ρυθμιστικά και μη ρυθμιστικά μέτρα την πλευρά της ζήτησης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα δεδομένου του μέγεθους της αγοράς μας να επηρεάσουμε τα πράγματα σημαντικά. Δεύτερον, έχουμε πολύ καλή εμπειρία τα τελευταία χρόνια δημιουργώντας πλατφόρμες ε, όπου συγκεντρώνονται πολλοί ενδιαφερόμενοι. Η κυκλική οικονομία είναι ένα καλό παράδειγμα το να έχουμε λοιπόν μια πλατφόρμα όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανταλλάσσουν και να αναπτύσσουν λύσεις που θα φέρουν αποτελέσματα για τα δάση, αλλά και που είναι και εφικτές και υλοποιήσιμες για τη βιομηχανία, για παράδειγμα, είναι μια σημαντική δεύτερη πρόταση που κάνουμε. Γνωρίζουμε το γεγονός ότι ε, και στον επιχειρηματικό κόσμο υπάρχει αναβρασμός ε, κυρίως με γνώμονα τους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να εντάξουμε την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις ε, υπεύθυνε επιχειρηματικές πρακτικές, εθελοντικές συμμετοχές και να λειτουργήσουμε και με συστήματα προτύπων και επιστοποίησης. Να τα ενισχύσουμε, να τα βελτιώσουμε, να τα κάνουμε πιο διαφανή και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στα πιστοποιητικά, στις πιστοποίησεις που παράγουν και τέλο, το ανέφερα και προηγουμένω, το 15% τη αποψήλωση των δασών σχετίζεται με την παρανόμη υλοτομία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το σχέδιο δράσης FLEGT και γι' αυτό έχουμε ένα νέο σχέδιο δράσης από το 2018 μέχρι το 2022 που εξετάζει το τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να υιοθετήσουμε. Αυτό επισημαίνει και το πόσο σημαντική είναι η αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού για την υλοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το EU Timber Regulation, που αφορά την εμπορική διάθεση ε, παράνομα υλοτομημένων προϊόντων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε επίσης και με τις διάφορες χώρες, ε, με τις χώρες εταίρους, ώστε να τις βοηθήσουμε να υλοποιήσουν μια αλυσίδα αξίας ε, που να προστατεύει τα δάση, να προωθήσουμε την σχετική οικονομία στις χώρες αυτές. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες ώστε να ενισχύσουν τις δικές τους, τα δικά τους ρυθμιστικά πλαίσια που προωθούν τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αποψήλωση των δασών δεν θα είναι απλά ένα ζήτημα που συζητούν οι. Ε, αρμόδιοι για το περιβάλλον, αλλά ότι θα συζητείτε στα υψηλότερα επίπεδα και θα υπάρχει σε όλες τις πολιτικές και τεχνικές συνομιλίες με τους εταίρους μας. Και επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε, όπως είπαμε, την, βελτίωση, την υποστήριξη για την διακυβέρνηση των δασών. None of this can be expected to happen. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να γίνει αν δεν υπάρξει αρκετή χρηματοδότηση. Εξετάζουμε λοιπόν διάφορου τομεί όπου θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε, να βοηθήσουμε να διοχετευτεί μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για τι βιώσιμε ε, δασικέ δραστηριότητε. Αυτό περιλαμβάνει διεθνή συνεργασία ε, σε οργανισμού ε, προϊόντων, αφορά την δημιουργία του σχεδίου δράσης για βιώσιμη χρηματοδότηση, συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και εμπορικές συμφωνίες. Θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο για την μάχη κατά τη αποψήλωσης των δασών, συμπεριλαμβάνοντας διατάξεις που αφορούν τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Τέλος, ο τελευταίο τομέα ε, στον οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η έρευνα και η καινοτομία προχωράμε με την ε, ίδρυση ενό παρατηρητηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποψήφιση των δασών και την υποβάθμιση των δασών. Θα μα βοηθήσει να παρακολουθούμε καλύτερα τι αλλαγέ ε, στη δασική κάλυψη παγκοσμίω και θα διευκολύνει και την πρόσβαση για όλου του ενδιαφερομένου και τι αναπτυσσόμενε χώρε ε, και τι χώρε παραγωγή και τι χώρε κατανάλωση, ώστε να βρίσκουν τα δεδομένα που χρειάζονται για να τα συμπεριλάβουν στι δράσει που θα υιοθετούν. Και τέλο, θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ε, παγκόσμιων και περιφερειακών συστημάτων πληροφοριών για να παρακολουθούμε τις ε, συνέπειες των δασικών πυρκαγιών. Αυτά λέει ουσιαστικά η ανακοίνωση. Θέλω να κλείσω με μια μικρή ε, επισκόπηση των επόμενων βημάτων. Αυτή τη στιγμή προγραμματίζουμε μια σχετικά μεγάλη διάσκεψη στην Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο για τα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τα διεθνή δάση προγραμματίζεται για τις 22 και 23 Ιανουαρίου του 2020. Προχωράμε με τη δημιουργία της πλατφόρμας ε, για το διάλογο μεταξύ ε, ενδιαφερομένων και κρατών μελών. Και δεν θέλουμε να χάσουμε άλλο χρόνο για την αξιολόγηση των επιπλέον ρυθμιστικών και μεριθμιστικών μέτρων ε, για την πλευρά της ζήτησης. Και επίσης ξεκινάμε με το ε, Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, και την Κομισιόν συζητήσει ε, για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου. Γιατί, όπω είπαμε, είναι επίγουσα η κατάσταση. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιμένουμε να ληφθούν τα μέτρα. Πρέπει να ξεκινήσουμε με την υλοποίηση ήδη από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. So... Ευχαριστούμε. Οπότε ανακοινώνεται ότι θα υπάρχουν ε, ρυθμιστικά μέτρα για τα επόμενα βήματα. Μετά την ομιλία δε της ε, κυρίας Φαντερ νομίζω ότι μπορούμε να ανεβάσουμε τον πύχη. Αυτό είναι και το πνεύμα της δικής μας Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν μια διαδικασία διάει τώρα. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο 8 ερωτήσεων. Πρωτού ξεκινήσουμε να καλωσορίσουμε μια ομάδα νέων ανθρώπων που κάθονται εδώ στα πίσω έδρανα από τη Γερμανία. Σας καλωσορίζω. Ναι, πρόκειται για μια τάξη από το σχολείο Ιωάννης Κομένιους από το Πίνερμπερκ της Βόρειας Γερμανίας και χαίρονται πάρα πολύ ε, γιατί αυτή η συζήτηση που έχουμε σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, ιδίως για τους νέους ανθρώπους. Ναι, λέει ο Πρόεδρος, και για το μέλλον μας. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ και τον Πεταλίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα εδώ και πολύ καιρό που αναδείχθηκε με επιτακτικότητα τις τελευταίες εβδομάδες και οι πολίτες πλέον απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό, αλλά και σε δύο εβδομάδες στην Ολομέλεια να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Συζητήσαμε χθε και στους συντονιστές και εγώ είμαι τη άποψη ότι το θέμα πρέπει πραγματικά να το χειριστούμε με συστηματικότερο τρόπο. Να διοργανώσουμε και μια ακρόαση, να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλία. Ε, Πίστηκα και από τα επιχειρήματα των άλλων συναδέλφων. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ούτε μπορούμε να επινοήσουμε κάποιες τέτοιες εύκολες και γρήγορες λύσεις. Χρειαζόμαστε αποτελεσματικές λύσεις που θα είναι μακροπρόθεσμες. Είχαμε κάποτε κάποια στιγμή και την ευκαιρία να κάνουμε κάποιες επαφές με βραζιλιάνους αξιωματούχους στη Βραζιλία, όπου ε, ένας ε, αξιωματούχος που δεν ανήκει στους υποστηρικτές του Μπολσονάρο μου είπε ότι ε, στη Βραζιλία η αίσθηση είναι πολύ διαφορετική Μπορεί κανείς να κάνει μια πτήση στην Βραζιλία, πεντάωρη, και να πετάει πάνω από δάσος μόνο. Επομένως είναι δύσκολο να πιστούν οι Βραζιλιάνοι ότι κινδυνεύουμε από την αποψήλωση των δασών όταν βλέπουν παντού γύρω τους δάση. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο να ε, αντιμετωπίσουμε την πολιτική του Μπολσονάρου, είναι πολύ ευρύτερο και πολύ βαθύτερο. Και βεβαίως αυτό συνδέεται και με το πώς ε, ε, χειριζόμαστε και διαχειριζόμαστε εμείς τα δικά μας δάση στην ε, Ευρώπη. Είναι και θέμα αξιοπιστίας. Πρέπει και εμείς να προστατεύσουμε τα δάση μας εδώ στην Ευρώπη, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες όπου τα δάση ε, στις χώρες μας υποφέρουν. Δεν θέλω να υπησέλθω σε περισσότερα θέματα ε, ούτε στο θέμα της συμφωνίας με τη Σουρ. Δεν θέλω να πω ότι ε, τα πάντα είναι τέλεια σε σχέση με αυτήν την ε, συμφωνία. Ούτε όμως θα ήθελα να την απορρίψουμε τη συμφωνία αυτή, διότι είναι και ένα εργαλείο για να επηρεάσουμε την πολιτική της κυβέρνησης της χώρας αυτής, των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε σε δύο άξονες. Φιλικότητα προς το περιβάλλον, αλλά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά υπενθυμίζω ότι έχει ο κάθε ομιλητή στην διάθεσή του για τον πρώτο γύρο. Η κυρία Αρένα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ για την ε, ανακοίνωση αυτή. γιατί ε, Εκεί περιλαμβάνονται δύο σημαντικές ε, Προτεραιότητε, καταρχάς να δουλέψουμε και την, κατά τη αποψήλωση και όχι μόνο για την αποψήλωση αλλά και σε ό,τι έχει και αφορά την κατανάλωση προϊόντων ε, του δάσους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και προτείνει μια πρωτοβουλία ε, ρυθμιστική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ενσωματώνει επίσης την οπτική του διεθνούς εμπορίου στο ζήτημα της ε, αποψήλωσης των δασών. Νομίζω λοιπόν πως είναι γενικά πολύ ε, σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Τώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την ανακοίνωση, ε, υποθέτω πως υπάρχουν κάποιες ιδέες για την ρύθμιση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τι είδου ρυθμίσεις θα μπορούσαμε να έχουμε. Ε, ε, κανονισμό, κανονισμό για το δάση έχουμε αυτή τη στιγμή αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε του ίδιου τύπου ε, ε ρυθμίσεις που αφορούν την έμεση αποψήλωση. Έπειτα μιλήσατε για συμφωνίες ελευθερών συναλλαγών. Εγώ συμφωνώ για το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε εμπορικές συμφωνίες με τα άλλα μέρη του κόσμου. Όμως αυτές οι εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να ενσωματώνουν όχι μόνο μια, όχι μια δεσμευτική μάλλον αξία ή τιμή για το περιβάλλον, αλλά και κυρώσεις. Γιατί δούμε τώρα τις ε, εμπορικές συμφωνίες μιλάνε για σεβασμό του περιβάλλοντος, συμφωνία του Παρισιού κτλ. Αλλά δεν προβλέπεται καμία, ε, είδους κύρωση σε τέτοιες εμπορικές συμφωνίες. Τι είδους κύρωση θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ώστε να μπορούμε να πούμε ότι αν δεν γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία, για, πούμε, μια χώρα παίρνει απόφαση να αποδασώσει τη χώρα, την ίδια της τη χώρα, όπως είδαμε στη Βραζιλία τι κυρώσει μπορούμε να επιβάλλουμε σε σχέση με τη χώρα με την οποία έχουμε υπογράψει. Ευχαριστώ πολύ. And, uh, uh, thank you to the Commission for the good work. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το εξαιρετικό της έργο. Σας διαβεβαιώ ότι η Επιτροπή μας θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να συμβάλλει, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη σημασία έχει το θέμα. Επίσης θέλω να τονίσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει μια πλειάδα χωρών όπου η διαχείριση των δασών είναι πλημελής, Βραζιλία, Καναδάς, τεράστιες πυρκαγιές πριν από κάποια χρόνια και δεν κατάφερε ο Καναδάς να τις σβήσει έγκαιρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Ρωσία, στη, Σιβηρία και ούτε εκεί φαίνεται να είναι ικανοί να τις ε, κατασβέσουν. Μετά υπάρχουν ε, και μια σειρά άλλες πτυχές. Ένα εκτάριο τροπικού δάσους έχει μεγαλύτερη βιοπικιλότητα από ολόκληρη τη Φιλανδία. Άρα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά τη σόγια, όπου η Ευρώπη είναι μεγάλος εισαγωγέας προϊόντων σόγιας και αυτό δεν είναι άσχετο με τα όσα συμβαίνουν στη Βραζιλία. Πρέπει να βρούμε λοιπόν ένα, μια λύση στο πρόβλημα αυτό. πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Να κάνω και ένα σχόλιο ε, για την, ε, για την ανακοίνωση. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πρωτοπόρος στο θέμα αυτό γιατί ε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο όρο αντί για το trailblazing που χρησιμοποιείτε, γιατί νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο καταλληλότερος. Κυρία Μέτζ, πυρκαγιές στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην ε, Ελλάδα, ακόμη και στη Σουηδία πέρσι. Και όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές, τα δάση δέχονται επίθεση, όπως για παράδειγμα ε, το δάσος του Αμαζονίου, που θυσιάζεται από τον Πολσονάρο για, την, για το λόμπι το αγροδιατραφικό. Χαίρομαι που η Κομισιόν αναγνωρίζει τη σημασία των δασών και συμμερίζεται τις ανησυχίες για, τις, για την πολύ κακή κατάσταση που βρίσκονται τα δάσκη. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στις προκλήσεις η ανακοινώση της Κομισιόν. Μιλάει η Κομισιόν για διάλογο και κίνητρα. Πρέπει εδώ και τώρα να θέσουμε ένα τέρμα στην αυτορύθμιση του κλάδου και να εισαγάγουμε δεσμευτικούς κανόνες. Πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες δεσμευτικούς υποχρεωτικούς για την κατανάλωση και τις εισαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Ευρώπη είναι μεγάλος εισαγωγέας κακάου, μεγάλος καταναλωτής ε, προϊόντων κρέατος και γαλακτικών προϊόντων. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε την συνεκτικότητα της πολιτικής μας. Ως παγκόσμιος εταίρος δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνάπτει συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με τον Μπολσονάρο που ανοιχτά καταστρέφει το δάσος του Αμαζονίου. Αυτό υποσκάπτει την ίδια τη θέση που θέλετε να κατακτήσετε. Στην ε, κατεξοδότηση πράξη που ε, ε, ε, θεσπίσατε, εντάξατε το φινικέλαιο, αλλά όχι τη, τη σόγια. Και μετά, γεωργία. 80% το, της αποψήλωσης των δασών οφείλεται στο γεγονό ότι θέλουν εκείνοι που την ε, πραγματοποιούν να μετατρέψουν τις εκτάσεις της δασικές σε καλλιεργόμενες εκτάσεις και ε, εκτάσεις εκτροφής ε, ζώων. Γι' αυτό και πρέπει να ε, μεταβιβάσουμε την χρηματοδότησή μας και να την ανακατευθύνουμε σε αγροοικολογικά project. Εγώ συγχαίρω την ε, την Κομισιόν για την ανακοίνωσή της, αλλά καλό να θεσπίσουμε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για την προστασία των δασών. Η κυρία Μπενιέ για το Άρντι. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι ανταλλαγές ε, οι εμπορικές ε, σημαίνουν ταυτόχρονα την προστασία όλων των ε, δασών. Είδαμε τι συνέβη με τον Αμαζόνιο φέτος και δεν πρόκειται μόνο για τον Αμαζόνιο και στην Μαύρη Αφρική αυτή τη στιγμή σοβούν πολλές φωτιές. Χρησιμοποιούν εκεί τις φωτιές για να κάψουν τις γης και πρέπει να δώσουμε τα απαραίτητα μέτρα. Εάν θέλουμε να σώσουμε τον Αμαζόνιο και τι δάσος του Αμαζονίου θα πρέπει να αποσυρθούμε από τις συμφωνίες όπως η Μερκοσούρ. Η αποψήλωση των δασών οφείλεται στην βούληση για δημιουργία νέων γεωργικών γεών. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρό το, ε, ναι, ε, ε, δεν συμφωνεί με αυτό και πρέπει εσείς να τον πείσετε. Επιπλέον τα υπερπόδια εδάφη δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Θα σας προτείνω να προστατέψετε και την Γαλλική Γουινέα που έχει σύνορα με τη Βραζιλία και που κινδυνεύει και αυτή από αποψήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Muchísimas gracias a la Comisión por la presentación de esta, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προστασία των δασών και της βιοπικιλότητας είναι κάτι κοινό ε, που μας αφορά όλους. Όλες οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται και εγώ ωστόσο θα ήμουν κατά αυτής της ε, απικιακού τύπου ε, ε, στάσης απέναντι στις χώρες εκτός της Ευρώπης. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που θέλει να καταστρέψει το δάσο τους, πιστεύω, ούτε και ο Μπολσονάρο που τόσο πολύ ε, αναφέρθηκε εδώ. Ε, πιστεύω πως υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να επαγρυπνούμε, αλλά κυρίως εδώ στο σπίτι μας. Εδώ είδαμε ότι η απόφαση της κυρίας Μέρκελ να κλείσει τα σπυρονικούς σταθμού είχε ως επίπτωση επίσης αύξηση των εκπομπών και κανείς δεν, δεν χαρακτηρίζει την κυρία Μέρκελ όπως χαρακτηρίζεται ο κύριος Μπολσονάρο. Ε, θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω πως υπάρχει πολλοί κόσμος που βρίσκεται πιο κοντά στο δάση. Εδώ η Επιτροπή, από ό,τι η Επιτροπή μας και οι Βρυξέλλες, πολλοί κόσμος κατοικεί μέσα στα δάση. Έχει ζήσει στην Ισπανία, ας πούμε, αιώνες μέσα στα δάση και ξέρουν και γνωρίζουν πώς να τα διατηρήσουν και πολλές, πολλοί κανόνες πολλές φορές είναι αντιπαραγωγικές, αφήνουν ε, ε, τα δάση τελικά απροστάτευτα, βο, βο, γεμίζουν από κλαδιά, από πούσια και πολλές φορές ξεσπάνε φωτιές πολύ ε, ξαφνικά. Ε, όπως επίσης ε, τα δάση, τα μεσογειακά δάση αλλά και η χαμηλή μεσογειακή βλάστηση είναι αυτά που ε, καλύπτουν κατά μεγαλύτερο κομμάτι την Ισπανία και την Πορτογαλία. Και αυτά τα εκμεταλλευόμαστε εδώ και πάρα πολλά αιώνες με πολύ λογικό και ισορροπημένο τρόπο και επωφελή τρόπο. Πιστεύω και εδώ έχουμε μία από τις περιπτώσεις όπου οι εξωτερικές παρεμβάσεις δεν ωφελούν. Ο πρόεδρο διακόπτη. Συγγνώμη, πρέπει όλοι να μείνουμε στα δύο λεπτά γιατί διαφορετικά δεν ε, ε, έχει νόημα, πιστεύω. Η κυρία Χάζεν κάποια ε, ο κόσμος φλέγεται πραγματικά. Παντού στον κόσμο βλέπουμε να καίγονται δάση, να αποψηλώνται τα δάση, να... στον Αμαζόνιο να καίγεται ο Αμαζόνιος και αλλά και στην Ευρώπη διάφορα δάση, στη Ρουμανία, στις κάτω Και οι συνέπειε είναι αισθητέ. Ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών βρίσκονται σε κίνδυνο εξαφάνιση. Πρέπει να προστατεύσουμε λοιπόν τα δάση μα. Πρέπει να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα. Ε, Συζητώντα όμω, ε, δεν οδηγούμαστε πουθενά. Θα πρέπει να αλλάξουμε το σημερινό γεωργικό μας σύστημα που οδηγεί στην εξαφάνιση φυτών και ζώων. Τι θα γίνει με το δάσος του Αμαζονίου στη Βραζιλία. Είναι αυτοφιές δάσος. Η καταστροφή δεν γίνεται μόνο εξαιτίας του Μπολσονάρο, αλλά και λόγω των δικών μας συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών. Κάθε χρόνο ε, εισάγουμε μισό εκατομμύριο ε, τόνος ε, σόγια και τεράστιες ποσότητες ε, βοηού κρέατος από τη Βραζιλία. Με άλλα λόγια, για το δικό μας κρέος και, κρέας και για το δικό μας ξύλο και για το Αμαζόνιος και τα πράγματα θα επιδεινωθούν εάν συνεχίσουμε την Συμφωνία Μερκοσούρ. Είναι ντροπή. Είναι εξωφρενικό που η κυρία Μάλμστρομ, η Επίτροπος Εμπορίου, αρνείται να έρθει εδώ να μας εξηγήσει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ελευθερών Συναλλαγών ο κύριος Βέλα ήρθε και μας εξήγησε τι κάνει και ποια θα είναι η προσέγγιση. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να ε, προωθήσουμε άλλους τρόπους διατροφής, να απομακρυνθούμε από την κατανάλωση κρέατος, από ε, να εγκαταλείψουμε ε, την εντατική κτηνοτροφία, να δράσουμε έτσι στην Ευρώπη ώστε να και να σταματήσουμε αυτή τη συμφωνία Μερκοσούρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Εύη από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που διαβάζω σε αυτή την ανακοίνωση της Επιτροπής ε, την έντονη αυτή επισήμανση των καταναλωτικών συνηθιών στην Ευρώπη. Δηλαδή, ε, τονίζουμε τις εισαγωγές που κάνει η Ευρώπη και που σχετίζονται άμεσα με την αποψηλώση των δασών. Ε, η έννοια αυτή της ολοκληρωμένης αποψήλωσης των δασών είναι απόρρια των δικών μας καταναλωτικών συνηθιών στην Ευρώπη για διάφορα προϊόντα που έχουμε ήδη αναφέρει. Ανέφεραν οι συνάδελφοι από τους σπόρους μέχρι τα ζώα. Αυτό έρχεται σε τεράστια αντίφαση όμως με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, όσον αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οπότε σας παρακαλώ πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε μια δράση πιο συνεχή, πιο συνεκτική, ε, πιο θαραλέα και πιο παγκόσμια. Πιο καθολική. Πρέπει να καταφέρουμε, όπω είπαν οι συναδέλφοι, να παρέμβουμε στι δικέ μα εμπορικέ πολιτικέ και στη δική μα κοινή γεωργική πολιτική με περισσότερο θάρρο. Και ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας πει διαβάζω. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που διαβάζω ότι υπάρχει μια απόπειρα επιτέλους να υπογραμμίσουμε και τη σπουδαιότητα ε, της κατανάλωσης κρέατος και να αναφερθούμε σε κάποια ισορροπημένη διατροφή. Ελπίζω επιτέλους να λάβουν θέση τα ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συστήσουν ε, μια σοβαρή μείωση της κατανάλωσης κρέατος στους Ευρωπαίους πολίτες. Και μια άλλη αντίφαση που διακρίνω είναι η εισαγωγή σπόρων που συχνά έχουν τροποποιηθεί γενετικά και η συνεχής έγκριση που συνεχίζει να δίνει αυτή η Επιτροπή σε γενετικώς τροποποιημένους σπόρους διάφορων ειδών χωρίς να λαμβάνει ποτέ υπόψη την αντίθετη άποψη του Κοινοβουλίου αυτού. Και επ' αυτού πιστεύω θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερες προσπάθειες και να λαμβάνει υπόψη τις αντιρρήσεις που γίνονται από αυτό εδώ το κοινοβούλιο για αυτό το θέμα, διότι να εισάγουμε σπόρους σημαίνει να αυξάνουμε την αποψήλωση στον υπόλοιπο κόσμο και πρέπει επιτέλους να πούμε ένα φτάνει. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν σας δώσω το λόγο, ενημερωτικά ε, ο Πέτερ Λίζε αναφέρθηκε στην ε, συνεδρίαση των συντονιστών χθες όπου η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων εκφράστηκε υπέρ μιας έκθεσης πρωτοβουλίας, ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας ε, σχετικά με την αποψήλωση των δασών. Μετά από την ανακοίνωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από τα όσα συνέβησαν φέτος το καλοκαίρι θα σας ε, κρατάμε ενήμερους όσον αφορά τη μορφή που θα έχει το πεδίο το αντικείμενο που θα καλύπτει αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία μετά από την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών σε περίπου 10 μέρες στο Στρασβούργο. Αλλά ήταν σημαντικό πιστεύω να το μοιραστώ μαζί σας στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης που ακριβώς είναι ε, ε, αφιερωμένη στην αποψήλωση που οφείλεται στις δικές μας εισαγωγές. Οπότε θεωρήσαμε ότι καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε εδώ το εργαλείο μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό το οποίο ε, καλύπτει η Κομισιόν και που θα διευκρινίσουμε, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς σε 10 μέρες περίπου. Δίνω το λόγο στην Κομισιόν για 5-10 λεπτά το πολύ, 5 λεπτά το πολύ, για να μπορέσουμε να έχουμε το δεύτερο γύρο ερωτήσεων στη συνέχεια. Yeah, thank you very Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ και για την υποστήριξη και για την επικοδομητική κριτική που ακούστηκε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κατά θέματα. Υπάρχει το ζήτημα της ε, ρύθμισης νομοθετικής, των μακροπρόθεσμων λύσεων, το ρόλο του εμπορίου, της αλλαγής στον τρόπο ζωής μας και η ανάγκη ε, ανάληψης πιο στοχευμένης δράσης. Θα προσπαθήσω με βάση αυτούς τους θεματικούς άξονες να ε, διαρθρώσω τις απαντήσεις που θα σας δώσω. Πολλοί τονίσατε ότι θα ήταν σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει μια ρυθμιστική προσέγγιση όσον αφορά τις εισαγωγές εμπορευμάτων που σχετίζονται με την αποψήλωση των δασών. Και βεβαίως δικαίως ε, απορείτε κι εσείς ε, και με ρωτάτε ε, τι μορφή θα μπορούσε να έχει ένας τέτοιος κανονισμός. Δυστυχώς θα σας απογοητεύσω, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε κάποια εικόνα, ούτε κάποια ιδέα για το τι είδους κανονισμό θα μπορούσαμε να προτείνουμε. Αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι θα αξιολογήσουμε τα ρυθμιστικά μέτρα ως προς την αποτελεσματικότητά τους και όπως είπε και ο Πρόεδρος, και σας το λέω και εγώ, η νέα Πρόεδρος της Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για την βιοπικιλότητα, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για την αποψήλωση των δασών. Για τα είδη των ε, κανόνων και των κανονισμών, και χωρίς να θέλω να προκαταλάβω οτιδήποτε θα ε, ήθελε ενδεχομένω η Κομισιόν να κάνει, γιατί είναι πολύ πρόημο αυτό, μπορώ να σα πω όμω ότι στην ανακοίνωση αυτή ε, η ανακοίνωση αυτή ε, βασίστηκε σε μια σειρά μελέτες που ε, διεξήγαμε και εξετάσαμε και τα διάφορα είδη νομοθετημάτων που θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε. Εξετάσαμε και το ζήτημα της δέουσας επιμέλειας και εσείς οι ίδιοι είπατε και το παράδειγμα της, ε, της καταπολέμησης της παράνομης υλοτομίας και της σχετικής οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε πράγματι να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο στο μέλλον. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εξετάσουμε κλαδικά μέτρα ή μια γενικότερη προσέγγιση. Αλλά όλα αυτά θα πρέπει να αξιολογηθούν ε, λεπτομερώς και πρέπει να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε ε, όλα τα στοιχεία σε επαφή με όλες τις χώρες ε, και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα, τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει ε, επίσης να έρθουμε σε επαφή και με τις επιχειρήσεις, γιατί δεν θα έχει νόημα να θεσπέσουμε μια εξαιρετική νομοθεσία η οποία δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί ή θα είναι πολύ δαπανηρό να εφαρμόζεται στην πράξη. Γι' αυτό και πολύ προσεκτικά αυτή τη στιγμή σας λέω ότι πρέπει σε πρώτη φάση να αξιολογήσουμε τις ε, διάφορες εναλλακτικέ ρυθμιστικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε και που θα μπορούσαν να αποβούν αποτελεσματικές στην καταπολέμηση της αποψήλωση. Επίσης, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες στον κόσμο θα πρέπει να ε, ε, καθοδηγήσουμε τους υπόλοιπους, ε, τις υπόλοιπες χώρες με το παράδειγμά μας. Και εδώ μπορούμε πραγματικά να ε, βασιστούμε στην, ε, στον κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας. Αυτό θα πρέπει βεβαίως να συνεχίσει να εφαρμόζεται. Πρέπει να εφαρμόσουμε την υπάρχουσα στρατηγική μας για τα δάση και με μεγάλο ενδιαφέρον έχουμε διαπιστώσει ότι πολλά κρατημέλη αλλά και πολλοί δήμοι μιλούν πλέον για την αποψήλωση, αποψήλωση βλέπουν ήδη τι αρνητικές επιπτώσεις έχει η κλιματική αλλαγή ε, στην καθημερινότητα των πολιτών και αυτό και θέλουν να αναλάβουν δράση για την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής, της αποψήλωσης των δασών. Η Γερμανία είναι, για παράδειγμα, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα ε, τέτοιων ιδεών που έχουν ε, κατατεθεί. Ε, μιλάμε δηλαδή για την αναδάσωση, για, για το φύτεμα νέων δέντρων στις πόλεις. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Φυσικά, ο ρόλος του εμπορίου είναι κρίσιμος στην συζήτηση για την αποψήλωση. Και αμφιβάλλω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ε, ε, για όλοι μας ε, για το τι ακριβώς είναι το, το εμπόριο. Μιλάμε πάντως σε κάθε περίπτωση για την εισαγωγή προϊόντων εδώ που σχετίζονται με την αποψήλωση των δασών. Όμως οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών είναι και ένα εργαλείο που έχουμε στα χέρια μα. γιατί ακριβώ μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε διάλογο με άλλε χώρε. Αν η συμφωνία με τη Μερκοσούρ κυρωθεί, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα δεσμεύεται και η Βραζιλία από τη Συμφωνία του Παρισιού. Τα κεφάλαια για τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντο είναι δεσμευτικά κεφάλαια σε αυτέ τι συμφωνίε και έχουμε και συγκεκριμένη διαδικασία ε, διαιτησίας. Βεβαίως, έχουν ειδικό χαρακτήρα αυτά τα κεφάλαια ακριβώς γιατί ε, περιλαμβάνουν και την κοινωνία των πολιτών και τον διάλογο. Και εδώ η κοινωνία των πολιτών πραγματικά ε, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Κάποιοι είπατε ότι πρέπει να δράσουμε δραστικά, ρηξικέλευτα και να κλείσουμε τι αγορέ μα για όλα τα εμπορεύματα που σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την αποψήλωση. Εμεί δεν συμμεριζόμαστε την θέση αυτή. Ε, αμφιβάλλω κιόλα αν κάτι τέτοιο θα ήταν συμβατό με του κανόνε του ΠΟΕ. Και επίση νομίζω ότι δεν είναι το είδο ε, των κανόνων ή μέτρων που ένας οργανισμός όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που ενα οργανισμο οπω η Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύει στη δύναμη του διαλόγου θα έπρεπε να πάρει. Εμείς ε, Αξιοποιούμε τη δύναμη της πυθούς. Όπως είπε και κάποιος συνάδελφος, ε, χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες λύσεις. Οι μακροπρόθεσμες λύσεις δεν μπορούν να είναι ποτέ η λύση που επιβάλλεις με τη βία σε άλλους. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον διάλογο και να πείσουμε τους συνομιλητές μας. Και εδώ το ζήτημα της αποψήλωσης ε, ε, φαίνεται ότι είναι επίσης ένα ζήτημα όπου πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές αυτές. Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Λοιπόν, περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Έχουμε έξι ευρωβουλευτέ που έχουν ζητήσει το λόγο. Αν έχουμε παραπάνω χρόνο, βεβαίω θα επιτρέψω και σε περισσότερου να πάρουν το λόγο. Αλλά σα παρακαλώ, ένα λεπτό ο καθένα. Η κυρία Νόβακ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίαση αυτή, την ανακοίνωση αυτή, την οποία διάβασα ε, με προσοχή. Όμως δεν βρήκα εκεί ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στη, Σλοβαν, στη Σλοβενία. Την ε, αποψήλωση των δασών που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές. Στη Σλοβενία είχαμε... Ε, είχαμε χιονόνερο ε, που για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που προκάλεσε σοβαρότατες ζημιές στα δάση μας. Δεν καταφέραμε δυστυχώς να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Ε, από την όλη κατάσταση ε, δυστυχώς βρήκαν γόνιμο έδαφος να πολλαπλασιαστούν ε, επιβλαβείς οργανισμοί που ξέρετε ότι δεν σταματούν και στα σύνορα. Δυστυχώς πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτή τη διάσταση του προβλήματος. Uh, Thank you. <laughs> Uh, I have a comment on a particular measure that is, is, is me, is my turn, isn't it? Uh. Βίζη, και εγώ είμαι, είναι η σειρά μου, εμένα είπατε. Εκτός μικροφώνου ομιλήτρια, δυστυχώς δεν ακούγεται. My one ear. Um, I'm curious to know just very shortly what is meant by regular... Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείται με τον όρο ρυθμιστικά μέτρα για την ενέσχυση των εργασιών για την καταπολέμηση της αποψήλωσης. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει. Όταν λέτε ότι πρέπει να υπάρχει και μια αξιολόγηση και μια ανάλυση. Γιατί καταλαβαίνουμε την ανυπομονησία που νιώθουν κάποιοι, αλλά πρέπει να είμαστε μετρημένοι ώστε να, να καταφέρουμε να ε, οδηγηθούμε σε λύσεις με χώρες ε, αναπτυσσόμενες. Το να χρησιμοποιήσουμε ε, ως όμοιρο τις εμπορικές μας συμφωνίες, αυτό θα ήταν λάθος. Αν θέλουμε να προωθήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη στις τρίτες χώρες, τι εννοείται λοιπόν με τον όρο ρυθμιστικά μέτρα και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει. Ευχαριστώ η κυρία Χόιτελαντ για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε την ε, κυρία Σουμέκερ, τη Διευθύντρια, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να εξασφαλίσουμε ότι θα εμποδίσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος, την αποψήλωση των ε, δασών, τις πυρκαγιές κτλ. Τα είπαν και οι συνάδελφοι. Θέλω όμως να τονίσω και τη σημασία που έχει η σωστή διαχείριση των δικών μας δασών και πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών. Και θέλω επίσης να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο Νίλ Στόρβαλτς, ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του, του κόσμου. Έχω και ένα ερώτημα για την Κομισιόν. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα τι κάνετε για να εξασφαλιστεί ότι οι εισαγωγές και η κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συμβάλλουν στην αποφύλωση των δασών σε τρίτες χώρες. Σας άκουσα να το αναφέρετε, το θέμα αυτό, όμως θέλω να μου δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα του πώς ε, εξυπηρετείται ο στόχος και όχι αυτά τα γενικόλογα μόνο που μας είπατε. Πρόεδρος διακόπτη την, ε, ε την ομιλήτρια η κυρία Ντέλη για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Δεδομένου ότι έχω ένα λεπτό θα μπω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Είναι ένα ζήτημα που σχετίζεται άμεσα με την κλιματική αλλαγή και να καταλαβαίνω ότι η Κομισιόν πρέπει να αξιολογήσει τα πράγματα και χρειάζεται χρόνο γι' αυτό, αλλά εμείς φυσικά ε, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και επίγουσα η κατάσταση. Ε, είπε η Κομισιόν ότι η κατανάλωση είναι το πρόβλημα, αλλά να πούμε πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν αν θέλει να δώσει κίνητρα για βιοκαύσιμα και άλλου είδους ε, βιοενέργεια, διαφορετικά για τα τρόφιμα, για τις ζωοτροφές, για τις καλλιέργειες, θέλει να όλα αυτά ε, να αντιμετωπιστούν που συμβάνουν στην αποψήλωση ε, των δασών και μιλήσατε για τι εμπορικέ συμφωνίε ω εργαλείο. Ανέφερε η Κομισιόν και τη χρηματοδότηση. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όλο ο κόσμο, αλλά είναι ηγέτιδα στην ανάληψη δράση ε, σε θέματα κλιματική αλλαγή. Πώ μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπογράφοντε τη Συμφωνία του Παρισιού που υποσχέθηκαν να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, για να προστατευτούν τα δάση, θα το κάνουν πράγματι. Ευχαριστώ κύριε Χόισλεν για τους πρασίνους. Συνάδελφοι, θα ήταν αφελές να ισχυριστεί κανείς ότι μπορούμε να πείσουμε τον κύριο Μπολσονάρο με επιχειρήματα να σταματήσει την αποψήλωση όταν υπογράφει συμφωνία που λέει ότι θέλω να αξιοποιήσω τον Αμαζόνιο, ε, τότε δεν πρέπει να απορρίσει κιόλα για το γεγονό ότι ξαφνικά εμφανίζονται πυρκαγιέ στον Αμαζόνιο για να ε, ε, χρησιμοποιηθούν οι δασικέ εκτάσει για την καλλιέργεια σόγια. Το ερώτημα είναι λοιπόν, η συμφωνία με τη Μερκοσούρ δεν περιλαμβάνει κανένα είδο κυρώσεων. Άρα είμαστε αναποτελεσματικοί. Το εργαλείο αυτό είναι αποτελε... αναποτελεσματικό. Και γι' αυτό ρωτάω την, την Κομισιόν. Είναι δεσμευτικό, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα αυτή η συμφωνία. Γιατί μου φαίνεται ότι δεν έχει. Επίσης, και στην Ευρώπη έχουμε ε, δάση που πλήττονται και απειλούνται. Στη Γερμανία ε, φέτος χάσαμε περίπου 100 εκτάρια δασών λόγω της ε, ξηρασίας, γι' αυτό και χρειάζονται, ε, χρειάζεται να ενισχυθούν επιχειρήσεις που ε, ε, καλλιεργούν δάση με αυτό το σκοπό, την αναδάσωση. Κύριος Βάλλας για την ΚΟΕ. Εκτός μικροφώνου, ο κύριος Βάλλας. Δεν ακούγεται εκτός μικροφώνου μιλητής. Your mic, please. So your name first and your mic second. <laughs> Το όνομά σας πρώτον και δεύτερον το μικρόφωνο σας. Η ευρεία συμφωνία για την προστασία και την ανανέωση των δασών ήταν δύσκολο να συμφιλειώσει τη θέση αυτή με τις εξελίξεις που έχουμε στη Συμφωνία Μερκοσούρ και στις υπάρξεις συμφωνίες γεωργίας με ε, χώρες παγκοσμίω. Διαφωνούμε ότι όλες αυτές οι πυρκαγιές ε, στον Αμαζόνιο ανοίγουν το δρόμο για καλλιέργειες που θα καταλήξουν σε, στα ράφια των σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Ε, όλοι οι μεγάλοι όμιλοι και οι πολυεθνικές ε, με διατροφικά προϊόντα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν συμμετέχουν σε όλα αυτά και δεν αποτελούν τροχοπέδι για μας για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και διαφωνείτε ότι αυτές ε, οι συμφωνίε, οι εμπορικέ συμφωνίε δεν κάνουν παρά να συνεχίζουν την εκμετάλλευση εκ μέρους της Ευρώπης ε, και τι γενοκτονίε που προκαλεί. Δυστυχώς αυτές είναι οι πραγματικές αξίε τη Ευρώπη. Ε, turn off your mic. Thank you. So, the two last questions we have the time to... Σας ευχαριστώ. Ήταν αυτές οι τελευταίες ερωτήσεις που έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε. Ο κύριος Γιζίκ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Έχω ένα πρακτικό μέτρο που πιστεύω ε, θα μπορούσε να καταπολεμήσει την αποψήλωση των δασών και αυτό είναι η φύτευση ενός νέου δάσους. Έπειτα, δεν, πρέπει να θυμίσουμε πως δεν φυτεύουμε δάση, αλλά δέντρα. Ε, βλέπουμε τι γίνεται με αυτά τα φυτεμένα δάση, τα δέντρα σπάνε, ε, ξεριζώνονται με τους ε, δυνατούς ανέμους. Δεν είναι κομμάτι ενός σταθερού ε, δάσους. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, πρέπει να το καταφέρουμε μέσω της αυστηρής προστασίας των υπαρχών των δασών και να επιτρέψουμε στα δάση να αναπτυχθούν μόνα τους και να δημιουργήσουν νέες περιοχές, δασικές περιοχές. Ε, πρέπει λοιπόν να μπορούμε να είμαστε κομμάτι της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ερώτηση, Μπόκχαρτ, από τους σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ. Έχουν απαντηθεί πολλά από τα θέματα στα οποία ήθελα να θέσω κι εγώ. Όμω αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και που το αναφέρει η ανακοίνωση είναι να ασκήσουμε την ίδια πίεση και στους ίδιους μας τους ε, εαυτούς. Γιατί η πυρκαγιά στον Αμαζόνιο δεν είναι άσχετη με την δική μας ε, κατανάλωση, με το δικό μας μοντέλο κατανάλωση και τις, και τις μας. Οπότε, θα πρέπει και στην ε, έκθεση που θα συντάξουμε, έκθεση πρωτοβουλίας, να αναφέρουμε και αυτό το ζήτημα της συμφωνίας με την Περκοσούρ. Όμως επίσης αυτό που με απασχολεί εμένα είναι πώς θα χειριστούμε το ζήτημα των αιθαγενών λαών. Πώς θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των ηθαγενών. Έχετε ως Κομισιόν ε, κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα μπορούσατε να μας περιγράψετε. Σας ευχαριστώ. Ε, θα ακούσουμε τις τελικές απαντήσεις ε, της Επιτροπής για το επόμενο πεντάλεπτο maximum. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν συμφωνείτε θα δώσω το λόγο πρώτο στη συνάδελφο από την DG DEFCO για κάποια ζητήματα που αφορούν ε, τα ε, οικονομικά. Μάλιστα, θέλουμε να τονίσουμε και τις ε, εξωτερικές πτυχές. Εμείς στην DEFCO εξετάζουμε το πώς μπορούμε να στηρίξουμε την αναπτυξιακή συνεργασία την βιώσιμη γεωργία και την βιώσιμη διαχείριση των δασών. Όπως ξέρετε, στην Προτείνεται ένας νέος κανονισμός για τη χρηματοδότηση των δασών, επίσης το EFST για τη χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση με τον ιδιωτικό τομέα. Εξετάζουμε λοιπόν ποια είναι τα μέσα που έχουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις από την Ευρώπη αλλά και από άλλες χώρες θα εξασφαλίσουν την βιώσιμη διαχείριση της ε, Γεωργίας. Να βοηθήσουμε δηλαδή τις χώρες ε, ε, εταίρους μας να αντιμετωπίσουν τις απάτες και να μην, να έχουν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη έτσι ώστε να μπορέσουν να, έχουν, να έχουμε συστήματα που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όμως ο κανονισμός είναι ακόμα υποσυζήτηση ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και μετά πρέπει να ξεκινήσουμε όλη την, ε, τον προγραμματισμό. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε και με τους εταίρους μας εκτός και για την επικοινωνία και υπάρχει ένα κομμάτι που αφορά τις εταιρικές σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα συνεχίσω από εκεί. Ε, ε, κατέγραψα το μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του κανονισμού. Έχουμε επαναλάβει ε, ποια, ποια είναι η δυνατότητα για κανονισμό και σωστά τονίσατε ότι αυτά τα αριθμιστικά μέτρα θα πρέπει να τα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, δεν θέλω να πω ότι μπορούμε να, μπορείτε να περιμένετε μια αριθμιστική λύση γρήγορα τώρα μέσα στο χρόνο. Αυτό δεν γίνεται γιατί θέλουμε να έχουμε μια ε, ορθή ε, πολιτική. Θα ήθελα να σας αναφέρω τις ε, συμφωνίες, ε, γιατί τις αναφέρατε και πάλι και εσείς. Να σας πω ότι οι εμπορικές συμφωνίες ε, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα τις έχουμε να συνοδεύονται από διατάξεις που είναι δεσμευτικές για τις χώρες εταίρους και σχετίζονται και με τη διαχείριση των δασών αλλά και για τη σεβασμό των ε, περιβαλλοντικών συμφωνιών και συγκεκριμένα της συμφωνίας του Παρισιού. Ξέρουμε ότι Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού υπάρχουν στόχοι και για να επιτευχθούν θα πρέπει να σταματήσει ε, η ε, αποψήλωση των δασών και να ισχύσει το μνημόνιο περί που ισχύει στη Βραζιλία. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι το Κοινοβούλιο εδώ και καιρό ανησυχεί για την αποτελεσματικότητα αυτών των εμπορικών συμφωνιών και ιδιαίτερα για την αποτελεσματικότητα του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης και του κατά πόσο μπορούμε αυτό να το ελέγξουμε μέσα αυτό το συμφωνίο. Συζητήθηκε και πάλι ε, αυτή τη βδομάδα μάλιστα ε, στην Επιτροπή Εμπορίου. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα κάναμε μια μακρά και επικοδομητική συζήτηση με τη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε όσον αφορά το, τα στοιχεία που ελέγχουμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα συμπεράσματα στα οποία φτάσαμε ήταν ότι όντως θα μπορούσαν να αναλυθούν και άλλα μέτρα ε, αναπερίπτωση και η Κομισιόν τόνισε πόσο σημαντικό είναι το να συνεχίσετε εσείς με την κράτη-μέλη να αναφέρεστε σε όλα αυτά να αναλύεται τη σημασία που έχει αυτό το σημείο για τις εμπορικές συμφωνίες και ότι η Κομισιόν συνεχίζει να εξετάζει διαρκώς αυτό ε, το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ και κατανοώ το έτοιμά σα. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και στα δύο θέματα και στην αποψήλωση των δασών και στο εμπορικό ζήτημα από την άλλη πλευρά. Ε, Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να ε, τηρείτε πάντα το χρόνο σας. Θα επανέλθουμε στα θέματα τα εμπορικά πολύ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την αποψήλωση και έχω καταλάβει ήδη πως δεν είναι η τελευταία η φορά που θα το συζητήσουμε γιατί έχει ε, μεγάλη σημασία. Προτείνω ένα-δύο λεπτά διάλειμμα και μετά περνάμε στο επόμενο σημείο.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 Je suis ravi d'accueillir. Euh, μου τον κύριο Πετισιονέ, που είναι Γενικός διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Κλίμα με τον οποίο θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, περί του ειδικού ζητήματος των κλιματικών αλλαγών ε, με τα όσα ήδη έχει προτείνει ο, η, η Κομισιόν αλλά και με ίσως και νέες ανακοινώσεις στις οποίες θα προβεί η, ο ή μέλλον πρόεδρος του Κομισιόν και το τι θα σημαίνει αυτό για τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050 για τη μείωση μειών 30 ή μειών 50% μέχρι το 2050. Νέοι ναι, σημαντικοί στόχοι από την Κομισιόν με βάση τα όσα έχουν ήδη γίνει και ε, όσον αφορά νέες πιθανές προοπτικές για την ε, υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων. Θα σας δώσω πρώτα το λόγο λοιπόν για 10-15 λεπτά και μετά θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω ότι σε αυτό το δεύτερο γύρο ανταλλαγή απόψεων θα μείνετε όλοι ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ. Εάν μου επιτρέπετε θα μιλήσω αγγλικά. Καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή να σας απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή σας, στη νέα σας σύσταση και ζητώ συγγνώμη από τον Αρία Σκανιέτε, εξ μάλλον μάλλον του Αρία Σκανιέτε, του Επιτρόπου που ταξιδεύει σήμερα. Θα ήθελα σύντομα να σας θυμίσω τι, ε, πού βρισκόμαστε και τι επιτύχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεύτερον, να πω στο βαθμό που μπορώ, σε μια κατάσταση που φαντάζομαι καταλαβαίνετε είναι κάπως περίπλοκη, για το τι θα κάνουμε στο νέα μας εντολή. Τρίτον, να τονίσω ότι παραλλήλως υπάρχουν συνέπειες ε, των όσων κάναμε την προηγούμενη εντολή που πρέπει να α, τα λάβουμε υπόψη. Και αυτό σημαίνει ότι... Ε, και μάλιστα μάλλον να σας δώσω και μια εικόνα γρήγορη, πολύ γρήγορη, των διεθνών μας δραστηριοτήτων. Λοιπόν, στη διάρκεια της περασμένης θητείας με την πολύ μεγάλη βοήθεια των προκατόχων σας εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που μας βοήθησαν να έχουμε πάντοτε μεγάλες φιλοδοξίες. Βλέπουμε επίσης στην εξέλιξη στη στάση του Συμβουλίου ε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Πολλοί από εσάς συμμετείχατε σε τριμερείς διαλογούς και γνωρίζετε πόσο ε, κοπιαστική είναι αυτή η διαδικασία. Και βεβαίως ξέρετε πολύ καλά πως ε, αυτά όλα δεν σταματούν στην προηγούμενη εντολή. Έχουμε την νομοθεσία που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε ε, θέση, δηλαδή μείον 40% εκπομπές μέχρι το 2030 και μάλιστα έχουμε και περισσότερα από αυτό εάν υλοποιηθεί σωστά η νομοθεσία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 θα φτάσει το 45% μείωση των εκπομπών. Και μάλιστα αυτή η νομοθεσία δημιουργεί το, τη βάση χωρίς την οποία θα, δεν θα ήταν δυνατή η περαιτέρω πρόοδος. Υπάρχει δηλαδή ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά το είδος, το βάθος και το εύρος της νομοθεσίας σε σύγκριση με τους στόχους 2030. Δεν είναι μόνο άλμα όσον αφορά τα νούμερα, αλλά και στο πώς έχουμε εμεί οργανωθεί και πώς αυτά θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και περισσότερο. Η μεταρρύθμιση δε έχει γίνει και λειτουργεί. Η μεταρρύθμιση σταθερότητας της αγοράς έχει εφαρμοστεί και η επόμενη φάση ξεκινά τον, του χρόνου και θα δούμε και είδαμε μάλλον ότι η τιμή του άνθρακα έχει αυξηθεί πάρα πολύ από ιστορικά χαμηλές τιμές. Η αγορά πήρε το μήνυμα, έχει προβλέψει τη μεταρρύθμιση και συνεχίζει να το κάνει αυτό με σταθερό τρόπο. Άρα λοιπόν όχι μόνο οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, αλλά η τάση συνεχίζει να είναι αυξητική, αλλά είναι μια πιο σταθερή ε, ε, ε, ανωδική πορεία, η οποία δίνει το μήνυμα προς την βιομηχανία του άνθρακα ότι πρέπει να προσαρμοστεί. Δύο λοιπόν στόχοι επιτυγχάνονται έτσι, περιβαλλοντική αικαιρεότητα και μείωση των εκπομπών. Μακάρι όλα να πάνε έτσι αίσια. Δεν υπάρχουν σημάδια ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Γιατί το τονίζω, γιατί χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσαμε καν να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα που είπε η ε, υποψήφια πρόεδρος της Κομισιόν όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική. Ριζικά αλλάζει η ποιότητα της νομοθετικής βάσης επί της οποίας θα στηριχθούμε για το μέλλον. Είναι ένα καλό παράδειγμα αυτό και από μια προσπάθεια μοιρασιάς της προσπάθειας έχουμε φτάσει σε έναν κανονισμό μοιρασιά της προσπάθειας που σημαίνει ότι η ε, τα κράτη-μέλη υιοθετούν αυτήν την υπόθεση. Έχουμε τον τομέα των γεών, ε, χρήση γεών, κατανομή γεών ε, και έχουμε επίσης τα στάνταρ για τα επιβατικά αυτοκίνητα αλλά και για τα φορτηγά έχουν ενισχυθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και έχουμε αυστηρότερους κανόνες και για τα βαρέα οχήματα όπου Αυτές οι προδιαγραφές βαραίνουν γιατί απαιτούν πραγματικές αποδείξεις και ε, ε, έχουμε βάσιμο λόγο να πιστεύουμε πως θα οδηγήσουν την αγορά προς τα καθαρά αυτοκίνητα. Ελπίζουμε ότι αυτό η ε, κίνηση θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να τα καταφέρουμε. Διαφορετικά θα χρειαστεί και άλλη μια γενιά στάνταρ ακόμα πιο αυστηρών και δεν θα διστάσουμε να προτείνουμε νέα στάνταρ. Ίσως ήδη έτσι να χρησιμοποιήσουμε την ρήτρα την, με ε, πρόθεσμης εξέτασης και αναθεώρησης. Πολύ σημαντικά λοιπόν πακέτο για το 2030 και φυσικά δεν χρειάζεται να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία ευαρέσκεια εδώ στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, στα κρατημέλη για το γεγονός ότι το 40 ή 45% αρκεί. δεν είναι νέα συζήτηση, είναι μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και καιρό και θα επανέλθω σε αυτό. Έχουμε επίσης ε, κάνει μέγα βήμα στην πρόταση του ανακοίνωση του περασμένου Νοεμβρίου με στόχο για το 2050, δηλαδή ουδετερότητα ε, κλιματική, μηδέν, ε, μηδενική ε, ανοχή μέχρι το 2050 και αυτό ήταν μέγα επιτεύγμα γιατί περικλεί τα όσα έχουμε κάνει παλιότερα. Δηλαδή στέλνει σαφές μήνυμα ότι τα πράγματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν, ε, οι πολιτικές έχουν σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ένας στόχος, αλλά ίσως όχι πια. Τώρα θα πρέπει να θέλουμε να πετύχουμε έναν ε, στόχο, αλλά με, το, με, με την σιγουριά ότι θα... Ε, αποκτήσει νέα διάσταση στο μέλλον, θα συνεχιστεί. Δηλαδή αυτοί οι στόχοι πληρούν έναν πολύ στρατηγικό στόχο που από τώρα δείχνει την επιρροή του. Και βέβαια αυτός ο στόχος δεν είναι ακόμα στόχος της Ένωσης, είναι πρόταση της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον ε, ε, ε, Ιούνιο δεν ήταν απόλυτα ικανοποιητικό. 24 κράτη-μέλη από τα 28 ήταν υπέρ και ε, ενώ τα τέσσερα μελη ζητούν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την εσωτερική συζήτηση ζητούν περισσότερη δουλειά για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε αυτή η στόχη να είναι ρεαλιστική. Δηλαδή, πού θα βρούμε τους πόρους βασικά για τις ε, μαζικές επενδύσεις που χρειάζονται για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτές τις αλλαγές. Το άλλο σημείο με το οποίο είμαστε πολύ ευχαριστημένοι είναι ότι Πώς επιθυμούσαμε τον περασμένο Νοέμβριο, αυτή η διαδικασία έγινε μέσω μιας πολύ ανοιχτή, διαφανούς και εντατικής συζήτησης σε όλα τα κρατημέλη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε αυτό, αλλά είδαμε ότι σχεδόν κανένα κράτος μέλος ε, μάλλον όλα τα κατεμέλια έκαναν την προσπάθεια να εξαπλώσουν τη συζήτηση μέχρι και στις περιφέρειες και στην ε, κοινωνία των πολιτών. Γιατί νομίζω πως αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί με τον αντίκτυπο που θα έχει στην κοινωνία μας πρέπει να χαίρει πολύ πολύ βαθιά συνένεση ε, από ολόκληρη την κοινωνία ώστε να μπορέσει να στηριχθεί τις επόμενες δεκαετίες. Πού βρισκόμαστε λοιπόν. Α, συγγνώμη και κάτι που ξέχασα και που είναι πολύ σημαντική καινοτομία είναι ο κανονισμός περί ε, διακυβέρνησης. Δεν είναι μια απλή γραφειοκρατική, ένα απλό γραφειοκρατικό πείραμα. Θέλουμε να φανεί η δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους μας, γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι ενώ η Ένωση πιθανότατα θα χρειαστεί και θα αντιμετωπίσει, θα φτάσει μάλλον τους στόχους 2030, ε, ε, θα υπάρχουν ε, εκπλήξεις ίσως, θα υπάρξουν προβλήματα που δεν τα έχουμε προβλέψει, τα νούμερα που δείχνουν ποια είναι η πραγματική τάση τα είχαμε στη διάθεσή μας πολύ αργά. Τώρα έχουμε όλα τα κρατημέλη με πολύ καλά σχέδια. Τα σχέδια αυτά τα έχουμε δει. Ορισμένοι, ορισμένα κενά είναι σημαντικά, ειδικά όσον αφορά την ε, επάρκεια σε ε, ενέργεια, αλλά δεν είναι και τόσο σημαντικά ώστε να είναι απαγορευτικά. Και έπειτα είμαστε ακόμα στο 2019 και άρα, άρα μέχρι το 2030 θα πρέπει να είναι δυνατό να διορθώσουμε αυτά τα προβλήματα. Ε, Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ο εντοπισμό των προβλημάτων εγκαίρω, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα και το χρόνο να τα διορθώσουμε, για να μην κάνουμε πασαλήματα την τελευταία στιγμή. Τώρα, πού θα πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και μετά. Είναι μια περίπλοκη κατάσταση για το Επίτροπο Φίσλερ, γιατί ε, επειδή ακόμα δεν έχει σχηματιστεί η νέα Επιτροπή, δεν ξέρω καν ποιος θα είναι το αφεντικό μου. Οπότε όχι, δεν το γνωρίζω ακόμα. Αυτή τη φορά έχουν κρατηθεί όλα εντυπωσιακά μυστικά. Δεν ακούσαμε καθόλου κουτσομπολιά. Αλλά μπορούμε να πούμε, καταλαβαίνοντας από τις πολιτικές ε, ε, κατευθύνσεις, ε, κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου Βαντερ Λάιεν. Σαφώς εδώ η Κομισιόν θα θελήσει να βασιστεί στο ακί, στο κεκτημένο και να κινηθεί γρηγορότερα από οποιονδήποτε άλλο παλιότερα. Θα υπάρξει δηλαδή, δηλαδή μια επιτάχυνση. Δεύτερον, κάτι που τονίζουν οι πολιτικές ε, κατευθυντήριες γραμμές είναι ότι τόσο η οικονομική και η πολιτική κατάσταση έχουν αλλάξει ε, ριζικά από το 2014 όταν ε, ήταν η τελευταία φορά που υιοθέτησε συμπεράσματα ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επ' αυτού και η Κομισιόν άρχισε να εργάζεται από αυτόν. Άρα λοιπόν η οικονομική μας ανάλυση είναι κάπως ξεπερασμένη. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα, ε, αλλά ήταν ε, πριν 4-5 χρόνια. Μετά ε, στηριαστήκαμε στη σύνταξη των ε, κανονισμών, έπειτα στην ανάλυση. Ε, οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν θέτουν το εξής ερώτημα, ότι αυτή τη στιγμή είναι ώρα να ξανασκεφτούμε αυτή την οικονομική ανάλυση όσο γίνεται πιο γρήγορα αλλά και όσο γίνεται πληρέστερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Ποια είναι δηλαδή η οικονομία που έχουμε ακριβώς ποια είναι η βάση για τις οικονομίες το 2019, ποια είναι η φιλοδοξία της Ένωσης που να μπορεί όμως να ε, ρεαλιστικά να επιτευχθεί μέχρι το 2030. Υπάρχουν και αρκετά πράγματα από τον οποίο έχουμε εργαστεί εντατικά τα τελευταία χρόνια, όπου μπορεί να μην είναι ο κατάλληλη στιγμή να μάλλον, ε, ε, συγγνώμη, μπορεί να είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε τι έχουμε καταφέρει εκεί. Ε, το σχέδιο βιώσιμων επενδύσεων που ξεκίνησε ο πρόεδρος Γιούνκερ μας δείχνει ότι το βασικό ζήτημα πίσω από όλα αυτά είναι μια μαζική προσπάθεια επενδυτική σε ολόκληρη την Ευρώπη για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτή είναι απόλυτη προϋπόθεση για αν θέλουμε να γίνει οτιδήποτε. Έχουμε δουλέψει για τη δημιουργία νέων και καλύτερων επενδυτικών εργαλείων. Έχουμε δουλέψει ώστε να ενταχθεί το κλίμα περισσότερο σε όλε τις γραμμέ του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Έχουμε δουλέψει ώστε να εξασφαλίσουμε πω ο υπόλοιπο προπολογισμό είναι σύμμορφο προ το Παρίσι. Και εδώ θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σα. επειδή εσεί πιέσατε πάρα πολύ για αυτό το ζήτημα. Ήταν κρίσιμη σημασία στο να γίνει αυτό. Κάναμε πάρα πολλή δουλειά όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Δημιουργήσαμε προϋποθέσεις πλαίσιο ώστε οι ε, επενδυτέ να γνωρίζουν αν και κατά πόσο η επένδυση είναι βιώσιμη ή όχι και όλα αυτά είναι σημαντικό να τα συμπυκνώσουμε σε ένα σχέδιο δράσης το οποίο να μπορεί να αλλάξει, να, με, να, να βελτιωθεί Έχουμε όμως στοιχεία για να μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα ε, πλάνο για βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης έχουμε τη στρατηγική μας ε, προσαρμογής που θα έχει θεωρηθεί πολύ επιτυχή, ενώ η προσαρμογή ε, θεωρεί το κάτι αδιάφορο. Ε, μόνο 10 κράτη-μέλη είχαν τέτοιο πλάνο προσαρμογής τώρα και 28 σχεδόν έχουν ολοκληρώσει αυτά τα σχέδια. Ανταλλαγή απόψεων, ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονικές γνώσεις έχουν πολλαπλασιαστεί. Έχουμε χάσει τον αριθμό το νούμερο το πόσα, το πόσα προγράμματα προσαρμογής των πόλεων υπάρχουν για την Κομισιόν πρέπει να προχωρήσουμε να, τώρα και να δώσουμε περισσότερη σάρκα στα οστά. Τώρα, ε, δουλεύουμε στην Κομισιόν για να εγκρίνουμε ένα σχέδιο για ευρωπαϊκές επενδύσεις για το κλίμα. Να δούμε επίσης, να συντάξουμε κατευθύντες γραμμές για το τι είδους προγράμματα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για να τεθούν σε διάθεση των αρχών, των τοπικών αρχών, των ασφαλιστικών ε, εταιριών, ώστε να μπορούν να ασφαλίσουν τις επενδύσεις αυτές. Ε, είναι λοιπόν σε μεγάλο βαθμό τοπικό θέμα αυτό, αλλά δεν είναι αδύνατο να συνδυάσουμε γνώσεις χρήσιμες ε, επαφές, χρήσιμες γνώσεις, ώστε να δούμε ποιο είδος κλίματος θέλουμε και ποια ε, σχέδια μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή να μπούμε στην προσαρμογή, στη στρατηγική προσαρμογή. Τρίτο σημείο εφαρμογή. Παράλληλα με τα όσα κάνουμε σε αυτή την εντολή όσον αφορά ε, τις νέες φιλοδοξίες είναι σαφές πως ε, η εφαρμογή των όσων έχουμε συμφωνήσει τα τελευταία πέντε χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Εάν δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε σωστή νομοθεσία είναι αυτοπάτητο να θεωρήσουμε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερες φιλοδοξίες. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο αυτά. Τέλος, η πρόεδρος Αντελάινερ σωστά τόνισε τις διεθνείς δραστηριότητες γιατί Αυτές ε, πολλαπλασιάζονται σε πελημερός και διμερός. Στην COP25 στο Σαντιάγκο θα έχουμε ένα πολύ βασικό ζήτημα. Ε, για να διαπραγματευτούμε. Όμως ε, παραμένει επίσης ε, ενισχύει το γεγονός ότι δεν θα δούμε τους εταίρους μας να ακολουθούν το δικό μας επίπεδο φιλοδοξίας εάν δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι εμείς το κάνουμε. Η χώρια μας στατηγική λοιπόν είναι το καλύτερό μας χαρτί όσον αφορά τη διεθνή δράση. Εάν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο οικονομικό και κοινωνικό το οποίο όλο ένα και περισσότερο είναι καθαρό και στο τέλος ουδέτερο κλιματικά και συνεχίζει να, δίνει, να προσφέρει ευημερία, τότε θα μπορέσουμε να πείσουμε τους, εταίρους μας, τους συνεταίρους μας να το ακολουθήσουν. Και υπάρχει μέγα ενδιαφέρον από πλευράς ε, αυτών των εταίρων, κυρίως από την Κίνα, να δουν τι κάνουμε, πώ το κάνουμε και αν τα καταφέρνουμε. Ευχαριστούμε για αυτή την πρώτη επισκόπηση του που βρισκόμαστε και την προοπτική του που θα πρέπει να βρεθούμε λογικά με την Επιτροπή. Ξεκινάμε με, την πρώτο, με τον πρώτο γύρο, δύο λεπτά ο καθένας μαζί με τους συντονιστές. Ξεκινάμε με το ΕΛΚΑ Πετρελίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Ναι, το ΕΛΚ υποστηρίζει τις προσπάθειες, ιδίως της κυρίας Φαντελάιεν, ε, για ενίσχυση της προστασίας του κλίματος. Άλλωστε έχουμε δεσμευτεί ε, να εξυπηρετήσουμε τον στόχο τη κλιματική ουδετερότητα. Όμω μα ενδιαφέρει πολύ αυτό που είπε η κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, ότι θέλουμε να έχουμε μαζί μα τον κόσμο, να προστατεύσουμε τι θέσει εργασία. και γι' αυτό ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο κύριο Γενικό Διευθυντή. Αν θέλουμε να είμαστε πρότυπο για τον κόσμο, τότε θα πρέπει και να συνεχίσουμε στην Ευρώπη να έχουμε βιομηχανία και θέσει εργασία στην βιομηχανία. Αλλιώ δεν πρόκειται να μα ε, ακολουθήσει κανεί. Εφαρμογή της ε, ισχύουσας νομοθεσίας. Είναι Πολύ σημαντικό αυτό. Θα ε, πρόσθετα δε ότι υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες ε, έχουν αποφασίσει να απαλλαγούν οι οικονομίες τους από τον ε, άνθρακα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο ETS. Συγκεκριμένα η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στην, στην αεροπλοεία. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, να υπενθυμίσετε και στους αδέλφους σας στην DG Move ε, ποια είναι η γραμμή της Κομισιόν, γιατί αυτά που ακούσαμε χθες ε, από τον συνάδελφό σας δεν μας πολύ Πρέπει λοιπόν να είμαστε σοβαροί και να μην ε, ισχυρολόμαστε ότι το Κόρζε ήταν κάποια φοβερή επιτυχία. Αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι σε ποιο, σε ποιο στάδιο της μετάβασης της ενεργειακής βρισκόμαστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό στην ε, διαδικασία αυτή να διασφαλίσουμε και τη διατήρηση της βιομηχανίας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές, ε, ε, κύριε κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε τον Γενικό Διευθυντή Πετριτσόνη που βρέθηκε μαζί μας εδώ σήμερα. Όπως είπατε, Πέρυσι η Ευρώπη πράγματι έλαβε μέτρα για να ενισχύσει με επιπλέον τις προσπάθειες μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών και για την ε, μετάβαση σε πιο βιώσιμη αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας. Αλλά δεν αρκούν αυτά, το ξέρουμε όλοι. Οι σημερινές προσπάθειες σίγουρα ε, καλύπτουν αρκετές από τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού και βοηθούν στο να επιτύχουμε την ε, μακροχρόνια, το μακροχρόνιο στόχο τη ε, κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Οι προσδοκίε τη νέα επιτροπή ε, και οι φιλοδοξίε είναι μεγάλε και παρατηρήσαμε και στο Κοινοβούλιο ότι η Ursula von der Leyen το είπε πολύ σαφώ ότι το κλίμα θα είναι προτεραιότητά τη κατά την θητεία τη. Αναμένουμε λοιπόν από την Κομισιόν να λειτουργήσει γρήγορα και αποφασιστικά και να βάλει την Ευρώπη στο σωστό δρόμο όσον αφορά το κλίμα. Αυτό πρέπει να γίνει και αποτελεσματικά. Ένας από τους καλύτερους τρόπους είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα ETS το οποίο θα διασφαλίσουμε ότι λειτουργεί σωστά. Είναι ο πιο αποτελεσματικός οικονομικά τρόπος ε, για να μειώσουμε τις εκπομπές στην Ευρώπη. Και θέλω να ρωτήσω την ε, Επιτροπή, σκέφτεστε να αυξήσετε την ετήσια ε, διάδοση του αποθέματος στην αγορά ώστε να μειωθούν οι εκπομπές. Και επειδή von der Leyen ανέφερε το ETS, και στο ναυτικό τομέα. Πότε θα δούμε να συμμετέχει ο ναυτικός τομέας, ο ναυτιλιακός τομέας στο ETS. Επίση, ε, όσον αφορά τον κανονισμό επιμερισμού των προσπαθειών, εάν η Κομισιόν σκέφτεται να χρησιμοποιήσει κάποια από την ευελιξία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη τη χρησιμοποιούν και αυτό δεν είναι καλό ε, για το κλίμα. Και τέλο, αναφέρατε τη νέα οικονομική ανάλυση που ε, επίκειται πότε ξέρετε, γιατί δεν θέλω να μας εμποδίσει από το να δράσουμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτές τις ε, ερωτήσεις, ε, πολύ σαφείς, για το Renew ο κύριος Στεφανούκα. Ευχαριστώ. Μιλώ εκ μέρους του συναδέλφου Νίλ Τόρβαλτς ε, και της ομάδας Renew Europa. Είμαι μέλος και της Επιτροπής Προπολογισμών. Αντιλαμβάνομαι κάποια γνωστική διχοτόμηση. Πριν το καλοκαίρι θέτουμε τεράστιους φιλόδοξους στόχους για τις εκπομπές και για το κλίμα και μετά το καλοκαίρι το Συμβούλιο ξαφνικά πάει να χρησιμοποιήσει χρήματα τα, αλλού τα οποία εμείς χρειαζόμαστε τόσο πολύ. Ήδη είναι δύσκολο να επιτύχουμε το 20% που αναφέρθηκε πριν από το καλοκαίρι. Η ίδια γνωστική ασυνέχεια ε, σχετίζεται και με τα κράτη-μέλη. Και η ερώτησή μου είναι πώ θα θέσουμε πιο δεσμευτικού στόχου στα κράτη-μέλη. Είναι θέμα διακυβέρνηση περισσότερο, όχι τεχνική ερώτηση, περισσότερο συνταγματική. Και τι εργαλεία σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για να γίνει αυτό, διότι σίγουρα δεν έχουμε κάποιο συνασπισμό ε, εθελοντών. Δεν είμαστε οι Ηνωμένε Πολιτείε όπου η Καλιφόρνια ε, έχει άλλους στόχους ε, από ότι το Ελληνό, για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει κοινέ στρατηγικές και κοινού στόχους. Ευχαριστούμε για τους πρασίνους, ε, Μισελ Μπλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που καταλάβατε και το ότι απαιτείται και δράση για το κλίμα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, ανανώσαμε το κοινοβούλιο και έχουμε ανανώσει και τη γενιά για το κλίμα. Στο δρόμο μας λένε ότι πρέπει να ακούμε τους επιστήμονες όταν δηλώνουμε και εμείς θεωρώ ότι έχουμε ευθύνη εδώ στο κοινοβούλιο για την επόμενη πενταετία να φέρουμε αποτελέσματα. Ο στόχος του 1,5 ε, βαθμού είναι ο στόχος. Ε, μόλις 60% είναι πιθανό να μην ε, μετατρέψουμε την γη σε θερμοκήπιο και να θερμανθεί η γη τόσο που να μην είναι κατοικήσιμη από ανθρώπινα όντα. Είναι μεγάλη πρόκληση. Οι ερωτήσεις που ακούσαμε τώρα ότι οι στόχοι του 2030 πρέπει να αυξηθούν. Εμείς θεωρούμε ότι και το 55% δεν είναι αρκετό. Τα σημερινά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια δεν βασίζονται σε αυτούς τους στόχους και εξακολουθεί να υπάρχει κενό. Τι θα κάνει η Κομισιόν μέχρι τα τέλη του έτους ε, για να συνοδέψει να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που να καλύψουν αυτό το κενό το οποίο όπως είπαμε δεν είναι αρκετό και επίσης εσείς ως Κομισιόν έχετε σκοπό να επιβάλλετε και δεσμευτικούς στόχους στο μέλλον αν τα κράτη-μέλη δεν καταφέρουν ε, να τα επιτύχουν όλα αυτά. Άκουσα τη σκέψη σας το τι άλλο μπορεί να γίνει. Μπορείτε να πείτε κάτι ακόμα για το, νομοθεσία για το κλίμα. Εμεί ε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μακροχρόνια στρατηγική και να αυξήσουμε του στόχου του 2030. Θέλουμε να υπάρχει ε, ένα ε, κλιματικό ολογισμό στην ομοθεσία, θεσπισμένο που να συνάδει με τη Συμφωνία του Παρισιού. Επίση, μιλήσατε για τα πρότυπα και την αναθεώρηση το 2023 και το 2020 και το 2023. Το ETS θα ξεκινήσει το 2021 η επόμενη φάση. Και ξέρετε, χρειαζόμαστε κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα. Είναι αναγκαίο να μειώνουμε κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα τις ε, εκπομπές μας. Μπορούμε λοιπόν από σήμερα να τροποποιήσουμε την τέταρτη φάση του ETS και επιβάλλοντας κάποιο ε, τιμή ε, για τον άνθρακα στο ETS. Ευχαριστώ, Σαρντόριν, για το ID. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο του ID. Πάμε στο ECR. Ο κύριο Βαντρά. Ευχαριστώ. Εδώ είναι το ECR. Παρόν. Είμαστε εδώ ως ε, συντηρητικοί για να εκπροσωπήσουμε όχι μόνο τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους ηλικία. Άμα θέλετε να επιτύχετε τους στόχους, ξέρετε ότι θα πρέπει να δώσετε κίνητρα στον κόσμο με καρότα, αλλά ακούσαμε πολλά και, αλλά ε, δεν ακούσαμε πολλά για τα μαστίγια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μιλάμε λοιπόν για ένα από τα τρία έγγραφο που θέλετε να συζητήσουμε με το λυρικό τίτλο «Δημοκρατική λήψη αποφάσεων προς μια Ευρώπη ε, πιο φιλική προς το περιβάλλον». Αυτό που εννοείται είναι βεβαίως η φορολογία. Νομίζω ότι είναι το χειρότερο τίτλος που έχω ακούσει ποτέ. Αυτό ο τίτλος ε, θα έπρεπε να είναι πώς θα ε, καταστρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παλιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απέφερε πλεονεκτήματα στους πολίτες της λόγω του ανταγωνισμού, ε, λόγω της ελευθερίας ε, κυκλοφορίας επιχειρήσεων. Γι' αυτό εμείς και εγώ και η χώρα μου προσχωρήσαμε στην, η χώρα μου προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τελικά καταλήξαμε να έχουμε δημιουργήσει έναν οργανισμό που στην ουσία απλά επιβάλλει φόρους από τα πάνω. Τώρα ακούμε και για κλιματικό περιβαλλοντικό φόρο είναι ε, κάτι το οποίο οδηγεί στη δραματική αύξηση το, της τιμής για τη στέγαση, για την ηλεκτρική ενέργεια, ε, ενέργεια. Πρόκειται για ανοιχτή πρόσκληση στους, ε, στα κίτρινα γελέκα ώστε να διαδηλώσουν σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Κομισιόν γνωρίζει τους κινδύνους μιας θέσπισης ενός τέτοιου ε, φόρου. Γι' αυτό και θέλει να συνοδεύσει τον φόρο αυτό από μέτρα ανακατανομής. Ε, εσείς ε, ε, ξέρετε, έχουμε εμπειρία στη χώρα μου από μεγάλες διαδηλώσεις. Δεν θα ήθελα να, να επαναληφθούν. Έχετε κάποιο σχέδιο ως Κομισιόν. Κάρας. Στο σχέδιο δράσης της Κομισιόν αναφέρεται ότι τα NECP θα πρέπει να ε, συμβάλλουν στην ολοκλήρωση υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο κύριος Γουάλλας μιλάει. Αυτή, αυτή, αυτές οι, αυτά τα σχέδια όμως περιλαμβάνουν και υποδομές ε, ε υδρορογμάτωσης που χρησιμοποιούνται ήδη στην, ε, στις ΗΠΑ. Ο Jean-Claude είπε στον πρόεδρο Τραμπ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να αποφύγει τους δασμούς στα αυτοκίνητα από τη ΣΥΠΑ, ότι θα αυξήσει την κατανάλωσή της αυτής της πολύ βρώμικης ρηπαρής ε, μορφής ενέργειας από την υδρορογμάτωση. Στην ε, Ιρλανδία η οικοδόμηση ενός τέτοι, μιας τέτοιας εγκατάστασης φυσικού αερίου, ορυκτού καυσίμου δηλαδή, ε, χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Κομισιόν. Το ερώτημά μου προς την Κομισιόν είναι, τι είναι πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη σας. Η εξασφάλιση της κερδοφορίας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας ή η εξασφάλιση της διατήρησης της ζωής στον πλανήτη. Δεύτερο ερώτημα. Πιστεύετε πραγματικά ότι είναι καλή ιδέα για την Ευρώπη να φέρνει σχιστολιθικό αέριο από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Πιστεύετε ότι πραγματικά αυτό είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον. Πρόεδρος, υπάρχει πλέον εκπρόσωπος ε, του ID στην αίθουσα. Όχι. Turn back to the, uh, the answers for, from the Commission for 7 uh, to 10 minutes. Ο εκπρόσωπος τη Κομισιόν έχει 10 λεπτά. Ναι, είναι δύσκολες οι ερωτήσει, αλλά θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Πρώτα απ' όλα, να υπενθυμίσω ότι η Κομισιόν ήταν πάρα πολύ σαφή. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική στρατηγική για το κλίμα, είναι η στρατηγική αυτή να είναι μια οικονομική στρατηγική. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση στην Ευρώπη, να διεξαγάγουμε τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες, αν δεν ε, είναι και μια στρατηγική για την ευημερία η στρατηγική αυτή. Και υπενθυμίζω ότι η οικονομία μας χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται επενδύσεις στον, ε, στον ε, βιομηχανικό μας μηχανισμό και εδώ ε, πρέπει να αποφασίσουμε, πρέπει να, να, να ακολουθήσουμε την πεπατημένη, δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα, ή θέλουμε να επενδύσουμε ε, χρήματα στις ε, καθαρές πηγές ενέργειας που θα κρίνουν και την κατάσταση του κλίματος τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτή είναι η θεμελιώδης ερώτηση στην οποία πρέπει να απαντήσουμε και αν δεν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα δεν θα έχουμε αποτελεσματική στρατηγική για το κλίμα. Θα κάνουμε διάφορα πράγματα αλλά δεν θα απαλλαγούμε από τον άνθρακα. Και αν δεν απαλλαγούμε εμείς στην Ευρώπη από τον άνθρακα δεν πρόκειται να, να το κάνει και κανείς άλλος στον κόσμο. Πρέπει να το επιτύχουμε για να αποδείξουμε ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο χωρίς να καταστρέψεις την οικονομία σου. Αυτός είναι και ο, η κεντρική ιδέα της στρατηγικής που πρότεινε πριν από λίγα χρόνια η Κομισιόν. Και πιστεύω ότι πρόκειται για μια πολιτική η οποία μπορεί να ε, επιτύχει τη συνένεση. Και αυτό είναι και το πνεύμα που θα διαπνεύσει όλες τις προτάσεις που θα υποβάλουμε από εδώ και στο εξή. Έγιναν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για το ETS. Φοβάμαι ότι σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη φάση, αν σας δώσω μια, την προσωπική μου γνώμη, θα σας παραπλανούσα, αν σας την έδινα. Πρέπει να προηγηθεί μια οικονομική ανάλυση η οικονομική ανάλυση στην οποία βασιζόμαστε αυτή τη στιγμή ε, έγινε πριν από πέντε χρόνια και τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βεβαίω θα χρειαστεί κάποιο χρόνο, δεν χρειάζεται όμω να περιμένουμε χρόνια και χρόνια. Από τη στιγμή που θα λάβουμε εντολή να ε, θα λάβουμε την εντολή να κάνουμε την ανάλυση, θα την ολοκληρώσουμε εντό ενό έτου. Και αυτή θα είναι η βάση για τι νομοθετικέ μα προτάσει. Και υπάρχουν πολλέ. Αναφέρετε κι εσεί κάποιε, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Όπω για παράδειγμα η αυστηροποίηση του ETS, όχι μόνο το αποθεματικό σταθερότητα τη αγορά, αλλά και η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων εκπομπών. Που ακόμα δεν έχει γίνει. Δεν έχουμε ε, δει ε, ποιε θα είναι οι θετικέ επιπτώσει των μειώσεων που ήδη έχουμε προβλέψει. Πιθανόν ε, θα πρέπει να αλλάξουμε το ETS προτού έρθουν και τα πρώτα καλά αποτελέσματα. Δυστυχώ έτσι είναι τα πράγματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε μια εις βάθος οικονομική ανάλυση για να έχουμε αξιόπιστα στοιχεία επί των οποίων θα βασίσουμε τις προτάσεις μας. Υπάρχει πρόταση για την παράταση του ETS και ε, την επέκταση του ETS. Η πρόεδρος ανέφερε την, ε, τον κλάδο των κατασκευών, της ναυσιπλοείας, της αεροπορίας όμω αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταργήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους τους ισχύοντες κανονισμούς και να φτιάξουμε καινούριου. Θα είναι μία από τις επιλογές που θα έχουμε στο τραπέζι, αλλά θα πρέπει κανείς να, να τα σταθμίσει όλα αυτά έναντι και των επιπτώσεων που θα έχουν. Η μόνη ευθύνη ε, για την ε, μείωση του ETS, των εκπομπών, θα είναι το ETS. Αν τον καταργήσουμε τον κανονισμό για τον επιμερισμό των βαρών, θα απαλλαγούν πλήρω τα κράτη-μέλη από τι ευθύνε του. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε αυτό. Δεν το ξέρω. Πρέπει να το σταθμίσουμε. Να το ζυγίσουμε και να δούμε. Πάντω, σε κάθε περίπτωση ε, θα ήταν ε, ανεύθυνο από πλευρά μα να σα υποβάλουμε ε, προτάσει χωρί να βασιζόμαστε να βασίζουμε τις προτάσεις μας αυτές σε πραγματική κατανόηση των πραγματικών δεδομένων. Σας είπα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε χρόνια και χρόνια. Εντός ενός έτους μπορούμε να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση αν μας δώσετε την, την ε, εντολή. Και από εκεί και πέρα να έχουμε στέρεες βάσεις για να υποβάλουμε τις προτάσεις που θέλουμε. Για τα ζητήματα που μου θέσατε σε σχέση με την προθυμία να προχωρήσουμε. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι εμείς θα προτείνουμε στη Νέα Κομισιόν να διεξαγάγει μια εις βάθος διαφανή οικονομική ανάλυση όλων των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας εντός του μικρότερου δυνατού χρονικού διαστήματος. Δίκαιη μετάβαση Ταμείο καινοτομία. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης εντάσσεται και συζητείται στο πλαίσιο του ΠΔΠ εγώ δεν συμμετέχω στι διαπραγματεύσει, μαθαίνω όμως από τους συναδέλφους και μπορώ να σας πω ότι ελπίζω ότι θα έχουμε ε, θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά για το MFF Φέτο και ότι εκεί θα εντάσσεται ένα ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο θα δούμε μια άλλη λύση, αλλά η δίκαιη μετάβαση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ε, βασικό στοιχείο του πακέτου. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι αν δεν αυξήσουμε τους πόρους μας και τα κονδύλια μας για τη δίκαιη μετάβαση και για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ε, με επιταχυμένους ρυθμούς, τότε ε, θα, αυταπατα, θα, θα πρόκειται περί αυταπάτης το να θεωρούμε ότι θα κάνουμε μια δίκαιη μετάβαση και μάλιστα ταχεία. Έως το 2030 χρειαζόμαστε πόρους για να εξασφαλίσουμε την ταχεία και δίκαιη ενεργειακή μετάβαση. Για το ζήτημα του προϋπολογισμού δεν ξέρω αν υπάρχει γνωστική ασυνέχεια ε, στην Κομισιόν. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Κομισιόν οφείλει να πάρει υπόψη της φαινόμενα και στοιχεία όπως είναι το Brexit, για παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή, ακούγοντας τις συζητήσεις στο Συμβούλιο, ε, βλέπω ότι υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στη φιλοδοξία που χρειάζεται περισσότερο ε, Περισσότερε επενδύσει γιατί πρόκειται για παραγωγικέ επενδύσει αφενός και αφετέρου την ε, απροθυμία να δοθούν και τα σχετικά κονδύλια. Αυτό δεν είναι ευθύνη της Κομισιόν. Ελπίζουμε παρόλα αυτά το τελικό αποτέλεσμα να μας δώσει τους πόρους που χρειαζόμαστε. NECP. Τα σχέδια αυτά ε, έχουν ως σκοπό τους να, δώσουν, να δώσουν την ευθύνη στα κράτη-μέλη, γιατί εκεί λαμβάνονται τα μέτρα. Έχουμε πει ότι αν σε τελική ανάλυση μέσω των ε, NCP, e τα κράτη-μέλη ε, δεν καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους που ε, περιλαμβάνονται στην νομοθετησία, δεν πρόκειται για δηλώσεις σκοπιμότητας πρόκειται για δεσμευτικά σχέδια τα οποία έχουν και υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η Κομισιόν θα προβεί και θα λάβει περισσότερα ε, μέτρα. Πάντω, ε, εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να τα πείσουμε ε, να βελτιώσουν και να καταρτήσουν αποτελεσματικά και σοβαρά σχέδια. Τα αποτελέσματα σε πολλές χώρες ε, τα, τα σχέδια στα οποία θα καταλήξουμε μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι θα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο που μα υπευλήθη έχουν αναλυφθεί σοβαρότατε πρωτοβουλίε. Στην Ιρλανδία, στι κάτω χώρε, έχουν ήδη γίνει αλλαγέ με τη βοήθεια τη Κομισιόν στα σχέδια αυτά. Θα είναι επαρκή όλα τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται σε αυτά τα σχέδια. Δεν μπορώ να σα το πω. Όμω, σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεκινήσει μια ει βάθο συνεργασία με τα κράτη-μέλη επί των σχεδίων αυτών, των NECP και νομίζω ότι θα έχουμε και επαρκή χρόνο στη διάθεσή μα για να παρακολουθήσουμε παρακολουθούμε και την υλοποίησή τους. Α, όλα αυτά τα στοιχεία θα υπάρχουν στην ε, ανάλυση, θα δημοσιευθούν και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Το μόνο που θέλω να πω ε, για τη φορολογία τώρα είναι ότι καμία περίπτωση σκοπός της Κομισιόν δεν είναι να καταστρέψει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, υποδομές φυσικού αερίου. Ας είμαστε ρεαλιστές. Τα ορυκτά καύσιμα δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τον κόσμο τα επόμενα χρόνια. Όμως υπάρχουν επιλογές και για το τώρα και για το μέλλον. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα στόχο για το 2050. Και γι' αυτό η κυρία Φόντερ Λάιεν ε, θέλει να καταστήσει αυτό το στόχο για το 2050 υποχρεωτικό. Αυτό που λέμε στην βιομηχανία και στον κλάδο του φυσικού αερίου είναι ότι ε, χαιρόμαστε που παρά το γεγονός ότι χαιρόμαστε ότι αντικαθιστούν το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή θέλουμε έως το 2050 να έχουν εξαφανιστεί και αυτοί από το μείγμα της ε, ενέργειας που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη. Μπορεί και να αποτύχουμε. Όμως ο στόχος που προτείνουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι να μην υπάρχει καθόλου διοξίδιο του άνθρακα έως το 2050 στην Ευρώπη. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δούμε όλες τις επιλογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπροστά μας. Όμως είναι σαφές, ο στόχος είναι πλήρης απαλλαγή από τον άνθρακα έως το 2050. Καθαρές μεταφορές, καθαρή κινητικότητα και γεωργικός τομέας, ο οποίος θα μπορεί να απορροφά όχι μόνο τις δικές του εκπομπές, αλλά και τις εκπομπές που προέρχονται από άλλους κλάδους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Ξεκινάμε με την κυρία Νταλή. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Θα εστιαστώ σε κάτι που μόλις ακούσαμε για τη συγχώνευση τομέων μεταφορές και οικοδομές στο ETS. Η συζήτηση αυτή έγινε πριν από πέντε χρόνια περίπου. Δεν έχω πιστεί ότι το αποτέλεσμα θα είναι καλό όταν μιλάμε ειδικά για τομείς όπως οι μεταφορές και οι οικοδομές και οι κατασκευές δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το τσιμέντο για παράδειγμα ή παρόμοιους τομείς όπως ο χάλιβας. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θα σας τα αναφέρω. Ρωτώ λοιπόν την Επιτροπή. Μπορούμε να μην βιαστούμε να βάλουμε τις οδικές μεταφορές και τις κατασκευές ε, στο ETS είπατε ότι θα ήταν πολύ βιαστικό, υπερβολικά βιαστικό να τα βάλουμε. Πρέπει πρώτα να εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία αξιολόγηση για το τι τιμή μπορεί να πετυχθεί για τι οδικέ μεταφορέ, για παράδειγμα, για να μην αναφέρω ότι πολλέ μελέτε τεκμηριώνουν ότι η τιμή ETS σε τέτοια περίπτωση θα ήταν αστρονομική και δεν θα κάνει κάποια διαφορά σε τομείς όπως οι μεταφορές. Γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε και εμείς ότι στοχευμένα μέτρα όπως τα πρότυπα ε, διοξίδιο του άνθρακα που επεξεργαζόμαστε είναι καλύτερα. Μπορούν να οδηγήσουν σε απαλλαγή από ανθρωπούχε εκπομπέ και να μα βοηθήσουν να επιτύχουμε του στόχου που ε, σε τελική ανάλυση θέλουμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε η κυρία Αρένα για τους σοσιαλιστές επίσης. Δεν υπάρχει επιπλέον ομιλητής από το ΕΛΚ, ε, Ευχαριστώ κύριε Πετριτσόνη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω εδώ ξανά στην Επιτροπή ΕΝΒΗ. Είχαμε συνεργαστεί παλιά στην ΙΝΤΑ. Η μείωση των εκπομπών μας ε, οφείλεται εν μέρη στην ε, μετατόπιση της παραγωγής ε, από την Ευρώπη στο πλαίσιο της απαλλαγής από ανθρακού εκπομπές στην ουδετερότητα ενεργειακά. Λαμβάνουμε υπόψη και αυτό. Αν λάβουμε υπόψη αν είχαμε όλη αυτή την παραγωγή στην Ευρώπη θα ήταν 30% αυξημένη η παραγωγή μας. Έχετε εισάγει αυτό το ζήτημα της δικής μας κατανάλωσης μέσω της μετατόπισης τη ε, παραγωγής. Δύο τομείς ε, θέλω να αναφέρω που ανέφερε η Μίριαμ, η σιδηρουργία και η χαλιβουργία συγγνώμη, και το τσιμέντο. Βλέπουμε ότι οι Ινδοί έχουν προχωρήσει περισσότερο από εμά σε θέματα πράσινη παραγωγή τσιμέντου ε, χωρί ανθρακούχε εκπομπέ. Ε, οι δικέ μα βιομηχανίε δεν έχουν επενδύσει σε νέε τεχνολογίε. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν τέτοιου τομεί ε, να επανέλθουν στι νέε τεχνολογίε για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί σε θέματα ε, ε, ουδετερότητα ω προ τον άνθρακα. Επανέρχομαι τώρα στην ε, Χαλιβουργία, όπου εκεί η Κίνα μα κάνει αθέμητο ανταγωνισμό ε, στι τιμέ και στι ανθρακούχε εκπομπέ. Εσείς Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει κάποια προσαρμογή ε, όσον αφορά τα θέματα των ανθρώπων εκπομπών. Η κυρία Σπυράκη για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτοιμη η Κομισιόν να ξανανοίξει το ETS, ε σωστά τα λέω ή όχι. Οπότε να σας ρωτήσω, ε, είστε έτοιμοι να προσθέσετε κάποιο μέτρα για συγκεκριμένους τομείς όπως τη μετοβιομηχανία και τη χαλιβουργία και αν φυσικά λαμβάνετε υπόψη τις ε, συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα και θέλω να μου πείτε και την άποψή σας για τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και που αφορά ε, το, το φόρο ε, για τους πρασίνους, ο κ. Πάρης. Um, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Γενική Διευθυντή. Ένα πράγμα δεν φαίνεται να είναι σαφές εδώ. Θέλω να κάνω μια επιστημονική δήλωση πρώτα απ' όλα. Βρισκόμαστε σε ε, επίγουσα κατάσταση για το κλίμα και απαιτούνται επίγοντα μέτρα. Και θέλω να μου πείτε, η οικονομική σας ανάλυση περιλαμβάνει και ανάλυση των ζημιών που θα Μα πλήξουν λόγω τη κλιματική αλλαγή. Όλοι βλέπουμε πλημμύρε καταιγίδε, ε, ξηρασίε ε, ε, που αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Αυτό θα επηρεάσει την οικονομία περισσότερο από ότι το κόστο που θα έχουμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. Υπάρχει κόσμο που αγωνίζεται για να επιβιώσει. Δεν πρόκειται να αγοράσει εισάγμενα πολυτελεία ευρωπαϊκά προϊόντα. Να είστε βέβαιοι και κάτι άλλο για το δικό σας φόρτο Να ξέρουμε ότι είναι μεγάλος και αυξάνεται. Όπως ξέρουμε, ε, η δική σας γενική διεύθυνση είναι σημαντικότερη από ποτέ αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να τα κάνετε όλα. Έχετε επαρκείς πόρους. Είναι, πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ε, lobbying για την Κομισιόν από τους Πρασίνους. Euh, Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, ε, κυρία Ριβαζή, από τους Πρασίνους. Κύριε Γενική Διευθύντα, αντίθετα από ό,τι λένε ορισμένοι συνάδελφοι, δείχνεται ότι η νομοθεσία για το κλίμα και την ενέργεια είναι εμβληματική η νομοθεσία της Ευρώπης. Εγώ υπήρξα εισηγήτρια για την ενεργειακή διακυβέρνηση και πρέπει να σας πω ότι το κείμενο με χαροποιεί από ευρωπαϊκής πλευράς, διότι είναι στρατηγικό το διακύβευμα. Ναι, τώρα λοιπόν έχουμε θέσει τους στόχους, αντιλαμβανόμαστε ότι οι στόχοι δεν βρίσκονται στο ύψος τη ε, ε, της COP21 και ότι χρειάζονται πιο φιλόδοξοι στόχοι, όπως είπατε πρέπει να, είμαστε, να δείξουμε μεγαλύτερη φιλοδοξία. Ταυτόχρονα, λέω, και θα ήθελα να μου απαντήσετε, για το 2020 Ποια κράτη δεν βρίσκονται στο ύψο των στόχων που έχουν τεθεί, αναρωτιέμαι. Μάλιστα, αν η Γαλλία έχει επιτύχει αυτού του στόχου του 2020. Έπειτα, είχαμε πει ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια στρατηγική για το μεθάνιο. Διότι το μεθάνιο επιβαρύνει πολύ τα αέρια θερμοκηπίου. Και ήταν η Κομισιόν να κάνει μια πρόταση σε σχέση με αυτό. Ε, τι συνέβη με αυτή την πρόταση. Και μετά, σε θέματα συνοχή, είπατε ότι η δική μα οικονομική ανάλυση είναι απερχαιωμένη. Εγώ βλέπω για το φυσικό αέριο. Προηγουμένω, ένα συνάδελφο μίλησε για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Ναι, τελειώνω. Αλλά και για τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών. Υπάρχει ε, ε, συνοχή όσον αφορά τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών, Μερκοσούρ, ΣΕΤΑ και την εθελοντική πολιτική όσον αφορά τα αερία θερμοκηπίου. Ευχαριστώ. Ο e. κύριος Κόκαλης από την ΚΟΕ. E. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Γενική Διευθυντά και ευχαριστούμε για το έργο σας. Υποστηρίζω την ιδέα των πρασίνων ότι έχετε την ε, πιο σημαντική γενική διεύθυνση στα χέρια σας ε, στην ιστορία του πλανήτη. Θέλω να θέσω το θέμα ε, των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων για τα ορεκτά καύσιμα δεδομένων των επενδύσεων που θα έχουμε στο μέλλον. Ακόμα επιδοτούμε σε πολλά κράτη-μέλη και με πολλές μορφές με φοροαπαλλαγές, τα εξωτερικά κόστη που ε, εσωτερικοποιούνται και έτσι στέλνουμε στην αγορά διαφορετικά μηνύματα αντί να φύγουν από τον άνθρακα. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για μια γρήγορη και σωστή μετάβαση των ε, περιοχών που θέλουν να εγκαταλείψουν τον άνθρακα και φτιάχνουμε ταυτόχρονα αντίστοιχα ταμεία. Ε, Πότε θεωρείτε ότι θα γίνει αυτή η μετάβαση για να κινηθούμε προς τους διανομής υγρών καυσίμων και τι θα γίνει με τις αδειοδοτήσεις ε, ε, για το πετρέλαιο στη Μεσόγειο. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, there were questions... Ευχαριστούμε. Ακούσαμε στον πρώτο γύρο ερωτήσει για την αεροπλοεία. Μπορείτε να την απαντήσετε ενδεχομένω από το ΕΛΚΑ για την κλιματική νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι προλάβατε ε, να απαντήσετε. Αν θέλετε, θα βρίσκεται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας φυσικά, οπότε θα θέλαμε μια απάντηση και επίσης χθες ε, είχαμε την ακρόαση της Κριστίν Λαγκαρντ ε, ενώπιον της Επιτροπής ΕΚΟΝ και θα έλεγα ότι το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο των ερωτήσεων αφορούσαν το ζήτημα του κλίματος και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κατά την άποψή μου έδωσε πολύ εθερετικές απαντήσεις. Η σύνδεση λοιπόν μεταξύ του δικού σας πακέτου, της δικής σας εργασίας, ε, ε, των καθημερινών σας εργασιών και των άλλων διευθύνσεων της Κομισιόν συμπεριλαμβανομένου του πακέτου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και πέραν της ε, Κομισιόν με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κάτι που εσείς θα πρέπει να έχετε στο νου σας και να σχολιάσετε ενδεχομένω την Επιτροπή μας. Αυτές ήταν οι τελευταίες ερωτήσεις. Έχετε 5-10 λεπτά για να δώσετε τις τελικές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Κυρία Άλλη, ε, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να δούμε τι κερδίζουμε αν βάλουμε στο ETS ε, τις μεταφορές και τις κατασκευές θα το εξετάσουμε. Ένα πράγμα για το οποίο είμαι απολύτω βέβαιο και μην το ξεχνάτε. Κοίταξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την επόμενη επιτροπή τώρα. Δεν είναι δικό μου ρόλο, ούτε μπορώ. Απλά θα προσπαθήσω να πω σαφώ ποιε είναι οι δικέ μου απόψει που θα χαρακτηρίζουν τι δικέ μου συμβουλέ προ την ε, Κομισιόν. Ε, αλλά κάτι που, για το οποίο είμαι απολύτω βέβαιο είναι ότι αν συμπεριλάβουμε τι μεταφορέ ε του ETS, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πρότυπα αυτή η κίνηση. Δεν θα, θα χρειαζόμαστε παρόλα αυτά ρυθμιστική δράση. Θα πρέπει να διατηρήσουμε και να υλοποιήσουμε τα πρότυπα διοξίδιου του άνθρακα για τις οδικές μεταφορές ούτως ή άλλως. Σε καμία περίπτωση δική, κατά δική μας γνώμη και των συναδέλφων μου δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτά που κάνουμε ήδη στον τομέα των οδικών μεταφορών με το ETS. Το κατά πόσο το ETS θα συμβάλλει επαρκώς στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές υπό όρους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα αλλού και να αξίζει τον κόπο δεν το ξέρω, θα το δούμε. Αν το αξίζει, αν αξίζει τον κόπο θα το προτείνουμε. Αν δεν αξίζει τον κόπο θα αναλάβουμε την ευθύνη και θα εξηγήσουμε γιατί δεν το προτείνουμε. Αλλά η στρατηγική που εθετήσαμε εμεί στον τομέα των οδικών μεταφορών, κατά την άποψή μου, είναι μια στρατηγική που πρέπει να συνεχιστεί και να υλοποιηθεί πλήρω. Και τώρα θα δούμε τι συμβαίνει με τα πρότυπα του 2020, γιατί συζητάμε για καιρό τώρα τα πρότυπα του 2030, αλλά του χρόνου θα δούμε πού βρισκόμαστε με τα πρότυπα του 2020, κατά πόσο έφεραν αποτέλεσμα στα προϊόντα που θέτουν στην αγορά οι κατασκευαστές μας. Είναι δύσκολο να απαντήσω ε, καθαρά στην ερώτηση τη κυρία Σαρένα και χαίρομαι μάλιστα που σας βλέπω και εγώ ξανά. Νομίζω ότι είμαστε όλοι ε, ε σύμμαχοι και ε, αντίπαλοι καμιά φορά κατά περίπτωση. Είναι κάτι που θα παρακολουθούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε εντάξει μέσα σε άκρες γιατί υπολογίζοντας τις επιδόσεις μας σε θέματα ε, κατανάλωσης και παραγωγής άνθρακα τα νούμερα είναι περίπου του ίδιου μεγέθους. Δεν εισάγουμε δηλαδή τεράστιες ποσότητες ε, περιεχομένου άνθρακα και σαφώς εξάγουμε λιγότερα προϊόντα άνθρακα. Αλλά αυτή είναι μια χονδρική εκτίμηση, ε, γενικευμένη. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Θα το συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε. Όσον αφορά το, η φορολογία, δύο πράγματα, διότι το φορολογικό ζήτημα ε, πολιτικά θα είναι ευαίσθητο. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το πολιτικό συμπέρασμα τελικά της Επιτροπής, αλλά η Πρόεδρος του είπε σαφέστατα, θα προτείνει τελωνιακή φορολογική ρύθμιση. Τι μορφή θα έχει δεν το γνωρίζω. Εγώ κοίταξα τις τελωνιακές φορολογικές ρυθμίσεις για άλλους λόγους, όλη μου την καριέρα στο εμπόριο. Ποτέ δεν απλοποίησα τα πράγματα. Επίσης υπάρχει και το θέμα των κινήτρων. Πολύ σαφές. Πόσο κίνδυνο είμαστε έτοιμοι να διατρέξουμε υιοθετώντα ένα μέτρο τέτοιου είδου ε, για να επιτύχουμε του κλιματικού στόχου. Αυτό είναι πολιτική κρίση, αλλά ο πρόεδρο τη Επιτροπής ε, ανακοίνωσε και πιστεύω εγώ δεν θα αλλάξει γνώμη ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Οπότε κάποια στιγμή θα προκύψει κάποια πρόταση, θα δούμε τι μορφή θα έχει και ποια θα είναι η συνέχεια. Η συνέχεια πιο γενικά πιστεύω παρότι δεν έχει λεφθεί καμία πολιτική απόφαση, πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε στενά την περιβαλλοντική φορολογία και την φορολογία του άνθρακα γενικότερα. Γνωρίζετε όλοι ότι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αγορά άνθρακα και όχι φορολογία άνθρακα ήταν διότι δεν θεωρήσαμε ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ποτέ στη φορολόγηση του άνθρακα. Τουλάχιστον έχουμε μία αγορά άνθρακα που λειτουργεί. Αλλά πολλά μπορούν να γίνουν. Το θέμα των επιδοτήσεων στα ορεκτά καύσιμα είναι θέμα φορολόγηση ουσιαστικά. Εγώ από τη δική μου θέση γνωρίζω πολύ καλά από την προηγούμενη δουλειά πόσο δύσκολο κάτι τέτοιο θα ήταν. Αλλά είναι παράλογο που δεν το εξετάζουμε καν ω ενδεχόμενο. Θα πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω με ποια μορφή. Δεν μπορώ να σα δώσω περισσότερε λεπτομέρειε γιατί ε, η συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα ε, μεγάλη ε, στην Επιτροπή και δεν ξέρω τι θα προκύψει από αυτήν, αλλά πιστεύω ότι και εγώ και οι υπόλοιποι συναδελφοί θα θέσουμε σε αυτό το ζήτημα ως ζήτημα το οποίο χρήζει εξέταση. Μερικές φορές για οικονομικούς λόγους, λόγω του πώς επηρεάζει την κλιματική πολιτική, άλλες φορές διότι είναι απλά δίκαιο. Μπορούμε να επιβαρύνουμε ορισμένα καύσιμα μόνο μέχρι ενό συγκεκριμένο ορίο σε σύγκριση με κάποια άλλη. Αλλά οι ζημιε από την κλιματική αλλαγή είναι σαφω Οι ζημιε από την κλιματική αλλαγή θα τι συμπεριλάβουμε ε, στην ανάλυση ε, για βάσει τη οποίε θα προκύψει μια στρατηγική προσαρμογή. Δεν χρειάζεται να είναι η ανάλυση για το ETS, αλλά στην πολιτική απόφαση αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, ε, τη μία προσπάθεια ή την άλλη, ή ει βάρο κάποιες άλλες για την απαλλαγή από τι εκπομπές. Φυσικά το βάρο των ζημιών πρέπει να ληφθεί υπόψη και ε, εσείς και το Συμβούλιο πρέπει να έχετε στα χέρια σα τα δεδομένα και εμεί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνεργαζόμαστε στενά με τον τομέα των ασφαλίσεων που του ενδιαφέρει ιδιαίτερα και παρόλα τα μέσα που έχουν και το προσωπικό που έχουν δεν ξέρουν για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς με κάτι θα πρέπει να, κάπου θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάτι ε, που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ούτω ώστε και εσείς και το Συμβούλιο να, μπορούμε να, να μπορείτε να αξιολογήσετε κατά πόσο αξίζει τον κόπο ε, το, η μία ή η αλλη τακτική για την απαλλαγή από τι ανθρακούχε εκπομπέ. Η στρατηγική αξία τη διακυβέρνηση, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ήταν ένα από τα καλύτερα νομοθετήματα και το βροντοφωνάζω. Γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί ούτω ή άλλω, οπότε δεν κατηγορώ κανένα, ούτε ευλογάω τα γένια μου. Ήταν πολύ καλό νομοθέτημα, περίπλοκο πολύ, γιατί είναι περίπλοκο το θέμα. Αλλά θα γίνουν εκτενείς προσπάθειες για καλύτερο σχεδιασμό. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος μίλησε επίσης για την ένταξη του κλίματος στο ευρωπαϊκό εξάμεινο κοιτάμε να δούμε πώς θα συντονίσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το εγχείρημα σχεδιασμού για τους διάφορους στόχους, για τα στρατηγικά σχέδια και οποιοδήποτε άλλο σχεδιασμό που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Πρέπει να επιτευχθεί κάποια ισορροπία μεταξύ του να σχεδιάζεις μέχρι θανάτου και του να ξέρεις τι κάνεις. Πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία. δίκαιη μετάβαση για τις ε, περιοχέ που παράγουν άνθρακα. Ναι, προτεραιότητα, αλλά όχι μόνο για αυτέ τι περιοχέ. Κάτι για τη δίκαιη μετάβαση. Το Ταμείο Δίκαιη μετάβαση είναι θεμελιώδη σημασία, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο εργαλείο. Το βασικό ερώτημα είναι το πώ θα δαπανίσουμε τα υπόλοιπα δημόσια χρήματα στην Ευρώπη. Είτε μιλάμε για ευρωπαϊκά, είτε για εθνικά. Η πολιτική συνοχή, η περιφερειακή πολιτική, είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αποσκοπεί στο να βοηθήσει ανθρώπους να μεταβούν από οικονομικά μη βιώσιμες δραστηριότητες κάπου αλλού. Πρέπει όμως να κάνουμε και πιο σκληρέ ερωτήσει. Πού θα τους πάμε. Διότι αν του τους πάμε σε μια άλλη δραστηριότητα η οποία σε 10 χρόνια θα αποδειχθεί να είναι μη βιώσιμη από κλιματική άποψη, σπαταλάμε τα χρήματά μα. Δεν είναι ριζοσπαστική αλλαγή, αλλά είναι μια σημαντική αλλαγή να ξέρουμε από πού ερχόμαστε, ξέρουμε ποιε είναι οι ευάλωτε περιοχέ, ξέρουμε ποια είναι τα ευάλωτα στοιχεία και οι ευάλωτε περιοχέ κατά κάποιο τρόπο με ελάχιστε. Ε, ε, ε, οι συνήθω ευάλωτε κλιματικά περιοχέ είναι και ευάλωτε οικονομικά. Οπότε τι κάνουμε με αυτέ τι περιοχέ, πού στέλνουμε τον κόσμο, ρισκάρουμε αυτού του εργαζομένου, για ποιο λόγο. Αυτό είναι βασικό και αφορά ολόκληρο τον προπολογισμό. Τόσο και όλου του προπολογισμού και τον ευρωπαϊκό και του εθνικούς και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτή την αρχή. Όσον αφορά το πετρέλαιο ως, When... ως ακινητοποιημένο περιουσιακό στοιχείο, ε, ναι, ε, δεν ξέρω το πότε. Δεν θα γίνει αν δεν έχουμε επαρκείς εγγύησεις για το πετρέλαιο. Τι κάνουμε λοιπόν, δημιουργούμε τις αγορές, τις τεχνολογίες για τις εναλλακτικέ πηγές και αυτό θα μας επιτρέψει να ξεφορτωθούμε και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Και πότε, το αργότερο σε 30 χρόνια. Νωρίτερα θα ήταν και καλύτερο. Ε, είναι δυνατόν, δεν το γνωρίζω. Ε, κλιματική νομοθεσία. Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας σίγουρα θα αποτελεί το επίκεντρο της κλιματικής νομοθεσίας οι στόχοι του 2030 δεν γνωρίζω. Θα είναι εντάξει τι είδους στόχοι 50-55 δεν θα το γνωρίζουμε τις πρώτες 100 ημέρες. Είναι πολιτική η απόφαση και ειλικρινά δεν νομίζω ότι μπορώ εγώ να δεσμευτώ αλλά θα αποτελέσουν κομμάτι της συζήτησης κατά πόσο είναι καλό ή όχι να έχουμε μια κλιματική νομοθεσία με στόχους του 2030, αλλά σίγουρα οι στόχοι του 2050 θα θέλαμε να περιλαμβάνουν μια σειρά αρχών που είναι κομμάτι της συλλογική μας δράσης στην Ευρώπη. Ε, κομμάτι από αυτά που προτείνει η Κομισιόν, τι ζητούν νομοθέτες, τι κάνουν νομοθέτες, ε, θέματα όπως μέτρα οικονομικής αποτελεσματικότητας, ε, θέματα όπως ε, δίκαιο, δίκαιος επιμερισμός βάρων μεταξύ κρατών μαλλών και κατηγοριών του πληθυσμού, της κοινωνίας, δίκαιη μετάβαση, η αρχή του να μην αφήσουμε κανένα να μείνει πίσω, αυτό το σλόγγαν να το κάνουμε νομοθεσία. Είναι δύσκολο. Κάποια τέτοια πράγματα θα θέλουμε αν μη τι άλλο να υπάρχουν στην κλιματική νομοθεσία για μένα, είναι δύσκολο να σα πω περισσότερα. Ξέρω ότι είναι γενικά αυτά που σα λέω και ότι δεν θα ικανοποιήσουν όλε τι απορίε, αλλά απαιτείται σοβαρή πολιτική συζήτηση στη νέα Κομισιόν πριν μπορέσουμε να πούμε κάτι πιο απτό. Οτιδήποτε και να σα πω άλλο θα είναι απλά προσωπικέ μου σκέψει. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε πίνοντα καφέ, αλλά δεν μπορώ σοβαρά να ε, ανακοινώσω τέτοια πράγματα εδώ σε αυτή τη συνεδρίαση βιώσιμη χρηματοδότηση και η σχέση με αυτά. Το μήνυμα της Προέδρου Βαντερλάιν νομίζω. Ξέρετε, ο Πρόεδρος Γιούνκερ υποστήριξε τη μακροχρόνια στρατηγική και την Ενεργειακή Ένωση. Η γραφειοκρατική διαδικασία, υπήρξε η γραφειοκρατική διαδικασία σε τελική ανάλυση θετική, η δουλειά έγινε. Το γεγονό ότι η νέα πρόεδρο λέει ότι θέλει το κλίμα να αποτελέσει βασική προτεραιότητα τη θητεία τη, το μήνυμα αυτό διευκολύνει τη γραφειοκρατική διαδικασία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά αν πάτε να δείτε την βιώσιμη χρηματοδότηση, σίγουρα θα έχετε ακούσει τον Ολιβιέ Γκεσά, ο οποίο, όπω ξέρετε, είναι η ψυχή του σχεδίου βιώσιμη χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών και ήδη έχει γίνει πολλή δουλειά εντός τη Κομισιόν χωρίς την οποία οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ε, δεν έχουν καμία σημασία. Η πρόεδρος ε, και η ομάδα της εργάστηκαν βάσει του κεκτημένου για την αεροπορία. Ξέρουμε ότι η αεροπορία είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα που έχουμε, διότι ακόμα δεν υπάρχει ε, σοβαρή τεχνολογική οδός προς την ουδετερότητα. Μπορούμε να παίξουμε με τα ηλεκτρικά αεροπλάνα, αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Τα εναλλακτικά καύσιμα, όσο και να πειραματοζόμαστε, το κατά πόσο θα βρούμε αρκετά βιοκαύσιμα για να λειτουργεί όλος ο στόλ, όλοι οι στόλοι όλο τον κόσμο χωρίς μαζικές ε, ε επιδράσεις στη χρήση γης, ε, είναι κάτι αδύνατον. Είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, σχετικά αποτελεσματική εφαρμογή εγχώρια με το ETS αλλά δεν πάει να είναι μεταφορά πόρων από την αεροπορία ε, στην απαλλαγή από ανθρακού και εκπομπές αλλού. Το μέσο αεροπορία σήμερα, πέραν των κερδών ε, της καλύτερης αποτελεσματικότητας, δεν έχει τα μέσα η αεροπορία για να προχωρήσει σε σοβαρή απαλλαγή από τι ανθρακούχε εκπομπέ. Είναι προτεραιότητα για μα στην Ευρώπη, διότι αυτό είναι ο ένα κλάδο όπου πραγματικά πρέπει να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, αλλά είναι δύσκολο αλλού μπορούμε να επιτύχουμε κάποιες ε, βελτιώσεις ε, εφαρμόζοντας κάποιους ε, πόρους. Η αεροπορία είναι ένα δυσκολότερο, ένας δυσκολότερος κλάδος. Αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέτε και εμείς έχουμε στην Ευρώπη μια αεροπορική βιομηχανία και όπως είπαμε το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τρόπο η βιομηχανία αυτή να υιοθετήσει κάποια αναλλακτική. Αυτό θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, να επενδύσουμε στην έρευνα για την αεροπορία, διότι χρειαζόμαστε ένα τεράστιο άλμα εκεί. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Για αυτήν την ε, εις βάθος ε, ε, εικόνα και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή και φυσικά θα περιμένουμε τις ακροάσεις με τον επόμενο επίτροπο ώστε να μπορέσουμε κάπως να τα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ένα λεπτό διάλειμμα και στη συνέχεια θα προβώ στις ανακοινώσεις του Προέδρου πριν το τελευταία σημεία για σήμερα. Okay, so we are going to Ωραία, λοιπόν, θα ξαναρχίσουμε στην ώρα μας ακριβώς. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας πάλι. ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις του Προέδρου σε σχέση με τις συστάσεις ε, των συντονιστών ε, από την συνεδρίαση της 22ης Ιουλίου. Οι συντονιστές σύστησαν και μάλλον οι συστάσεις αυτές έχουν κυκλοφορήσει ηλεκτρονικά. Φαντάζομαι δεν υπάρχει αντίρρηση, οπότε μπορούν να εγκριθούν. Οι ε, συστάσεις της χθεσινής συνεδρίασης θα κυκλοφορήσουν επίσης ηλεκτρονικά όσο γίνεται πιο ε, σύντομα, αλλά θα ήθελα να τονίσω κάποιες από τις ε, συστάσεις από τη χθεσινή μας συνεδρίαση γιατί θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε καιρός από πολιτική άποψη και όχι μόνο από διαδικαστική. Η πρώτη λοιπόν είναι ότι μετά από την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε χθε. για το Κόρσια, οι περισσότεροι αποφάσισαν ε, ε, να στείλουμε δύο επιστολές, μια προς το Συμβούλιο και μια προς την Επιστελή, για να τους καλέσουν να λάβουν πρωτοβουλία. Γιατί εχθές ανέλαβε τη θέση της για το Κόρσια η ε, Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο της 20 Σεπτεμβρίου θα το ε, αποφασίσει. Η πλειοψηφία λοιπόν αποφάσισε να στείλει μια επιστολή όπου θυμίζουμε τις ανησυχίες μας για τις πιθανές απειλές, το, αν το ETS ε καλύψει και την αεροπλοεία και λόγω αυτής της ε, γλώσσας αποκλειστικότητας ε, του ψηφίσματος για το Κόρσια. ξεκολουθούμε λοιπόν να πιέζουμε όχι μόνο την Επιτροπή αλλά και άμεσα το Συμβούλιο και φυσικά θα σας ενημερώνουμε για την αντίδραση του Συμβουλίου μέχρι να, τη συνεδρίαση της 28ης ε, ε, Σεπτεμβρίου. Επίσης, αποφασίσαμε να καλέσουμε την Επίτροπο Μάλμστρομ για το Μέρκοσουρ και είχαμε ανερνητική απάντηση από την Επιτροπή Μάλμστρομ ε, για λόγους χρονοδιαγράμματος. Θεωρήσαμε ότι οι λόγοι χρονοδιαγράμματος δεν μπορούν να αποτελούν το λόγο για να σταματήσει κανείς αυτό, αυτό και σίγουρα χρειάζεται συζήτηση με την Επίτροπο Εμπορίου ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου και βεβαίως θα στείλουμε νέα ε, πρόσκληση και θα επιμείνουμε περί της πολιτικής βούλησης της Επιτροπής μας ώστε να γίνει η ανταλλαγή απόψεων με, τον με την Επίτροπο Εμπορίου Τρίτο θέμα είναι τα γραπτά ερωτηματολόγια για τις ακροάσεις. Όπως ξέρετε, για τις ακροάσεις των νέων επιτρόπων θα έχουμε προφορικές ερωτήσεις και απαντήσεις, ε, αλλά και γραπτές ερωτήσεις και απαντήσεις. Οπότε ε, θα πρέπει να λάβουμε την απόφαση στην Επιτροπή ότι εσείς οι εκπρόσωποι θα, ε, δώσετε στους συντονιστές την αρμοδιότητα για να συμφωνήσουν για τις γραπτές απαντήσεις. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για τη γραπτή ε, διαδικασία. Εμείς θέλουμε λοιπόν την επίσημη έγκριση ώστε να συντονιστεί η, η, αυτά τα θέματα. Φαντάζομαι να μην έχετε αντίρρηση γι' αυτό. Οπότε οι συντονιστές πολύ σύντομα λοιπόν θα συντάξουν και θα συμφωνήσουν επί των γραπτών ερωτήσεων και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να ε, εσείς θα έχετε την ευκαιρία να θέσετε τις ερωτήσεις προφορικά στη διάρκεια της ακρόασης. Αυτές είναι οι συστάσεις λοιπόν που προέκυψαν από τη χθεσινή συνεδρίαση. Θα δούμε και άλλες για την αποψήλωση των δασών και ούτω καθεξής, αλλά φυσικά σεβόμαστε τη διαδικασία ενημέρωσης. Και τώρα θα περάσουμε στην τελευταία ανταλλαγή απόψεων που έγινε σήμερα το πρωί για την ε, έκθεση 2019 για την περιβαλλοντική εφαρμογή σχετίζεται με τα χθεσινά. Δεν, έχουμε να, θέλουμε μόνο να θεσπίζουμε στόχους, αλλά και να εφαρμόζουμε πολιτικές. Και για πρώτη φορά έχουμε αυτή την ανάλυση από την Επιτροπή για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά την εφαρμογή της κλιματικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Είναι καλό να έχουμε λεπτομερείς ε, παρουσιάσεις και ανακοινώσεις από την Επιτροπή και αυτό θα κάνουμε τώρα θα καλέσω τον, την κυρία Δωροθέα Σουμπάνου ε, να πάρει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση αυτής της αναλύσεως. Τον κύριο Σουμπάνου Δωροθέα, λοιπόν. Ε, καλησπέρα σας, ε, καλημέρα σας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το χρόνο και για αυτή τη συζήτηση και για τη συζήτηση της ε, έκθεσης ε, ε, περιβαλλοντικής εφαρμογής που είναι μάλιστα ο δεύτερος, δεύτερη φορά δεύτερη φορά που η Κομισιόν εκπονεί τέτοια έκθεση. Εγκρίθηκε τον Απρίλιο από την, το σύλλογο το σύνολο της Επιτροπής και θα ήθελα να σας καλέσω να δείτε το δίκτυο, το ιστότοπο αυτής της Επιτροπής που γίνεται εκεί ε, με την Γραμματεία και είδαμε ότι η οριζόντια εφαρμογή της Κομισιόν έχει τοποθετηθεί στο, το ιστότοπο, αλλά θα σας ε, καλούσα θερμά να δείτε και τις εκθέσεις των χωρών, διότι δεν είναι μόνο η οριζόντια επικοινωνία, η επικοινωνία, δηλαδή ο εντοπισμός των τάσεων, όσον αφορά τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις στον Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό ε, Νόμο, αλλά έχουμε εξετάσει με πιο πολιτική χρειά σε ποια κατάσταση βρίσκεται κάθε χώρα στους διάφορους τομείς, νερό, διαχείριση αποβλήτων, αέρας, βιοποικιλότητα, κυβέρνηση του περιβάλλοντος. Έχουμε εξετάσει όλα αυτά γιατί ε, ε, Είχατε και προσκεκλημένο τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης για το Κλίμα. Εξετάσαμε τη συσχέτιση ανάμεσα στην περιβαλλοντική πολιτική και την κλιματική πολιτική γιατί όπως ξέρετε υπάρχουν αντιστοιχίες και επιρροές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Επίσης εξετάσαμε την πλήρωση των διεθνών μας υποχρεώσεων που τις έχει αναλάβει όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά ως μέλος της Ένωσης. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε, γιατί είναι πολύ αλήθεια και μην διστάσετε στην παρουσίασή σας να εστιάσετε και να τονίσετε κάποιες εθνικές καταστάσεις. Μάλιστα, μάλιστα κύριε Πρόεδρε, θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι για δεύτερη φορά, όπως έλεγα, η παρουσίαση αυτού, αυτής της έκθεσης εφαρμογής. Έχουμε ένα σύνολο αναλύσεων και ποιος είναι ο στόχος. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, είναι σημαντικό όχι μόνο να αριθμίζουμε για τους πολίτες, αλλά και για την οικονομικούς φορείς είναι σημαντικό και πιστεύουμε και για την διεθνή φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ε, αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα μάτια των πολιτών, να έχουμε και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Ε, να τα δείχνουμε κιόλα στη στιγμή που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν υιοθετήσει νομοθεσία κάποιες φορές 10-15 χρόνια πριν και αυτή η, από, η νομοθεσία δεν έχει δώσει ε, ακόμα καρπούς. Αυτό το είδους ανάλυση γίνεται για να σας προσφέρει να προσφέρει και στους πολιτικούς, στους ευρωβουλευτές και βουλευτές στην Ένωση πιο πολιτική χρειά, ε, οπτική όχι προκατελημένη ε, εικόνα, αλλά μια γενική εικόνα ε, για την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να περάσετε και να διαβάσετε διάφορες διοικητικές εκθέσεις ε, που προετοιμάζει η Κομισιόν για την αξιολόγηση της τάδε της οδηγίας. Αλλά Εκεί δεν μιλάμε τόσο ξεκάθαρα για την κατάσταση των κρατών μελών, ενώ εδώ σε έχετε, εδώ σε αυτήν εδώ έχετε την κατάσταση σε διάφορους τομείς στα κάτι μελη και τα απορίσματα είναι σαφή και μπορείτε να τα βρείτε στις τελευταίες δύο σελίδες της οριζόντιας ανακοίνωσης. Έχουμε πολύ φιλόδοξους, φιλόδοξη περιβαλλοντική νομοθεσία ε, στην Ένωση, ίσως την πιο φιλόδοξη σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουμε σημαντικά επιτάγματα το ε, νερό της υδατοδότησης είναι ασφαλές, είναι πόσιμο στις περισσότερες αστικές και ε, περιοχές και περιοχές υπέθρου. υπαίθρου. Έχουμε κάνει καλή πρόοδο προς πιο κυκλική οικονομία. Πριν από τέσσερα χρόνια ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι θα απαγορευόταν η χρήση ε, ε, πλαστικών μιας χρήσης. Το καταφέραμε και αυτό, αλλά κυρίως με τα στοιχεία και τις στατιστικές και σας καλώ και πάλι να δείτε τις κατά χώρα εκθέσεις αναφορές ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές προκλήσεις ανάμεσα στα βασικά πορίσματα. Η πρόληψη των ε, αποβλήτων είναι σημαντική πρόκληση. Νέα χώρες τα πάνε καλά και πέντε έχουν ήδη φτάσει στους στόχους ανακύκλωσης που ορίζονται για τον επόμενο χρόνο, αλλά 14 κατημέλη κινδυνεύουν να χάσουν τους στόχους, οπότε μόνο ένας χρόνος μένει, λιγότερο από ένας χρόνος, μέχρι το 20. Ε, στην μισή Ευρώπη λοιπόν οι στόχοι ανακύκλωσης μπορεί και να μην επιτευχθούν. Για την ποιότητα του αέρα 18 κάτι μελη πάνω από τα μισά, Πρόεδρε, ε, προσπαθούν ε, με το οξύδιο του αζότου ε, Επίσης, ε, έξι έχουν προβλήματα με τα, με τα μικρά σκοματίδια, τα 10 ε, και 2,5 που είναι πολύ επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Τα περισσότερα ακόμα πασχίζουν να ολοκληρώσουν το δίκτυο Natura 2000 ε, των προστατευόμενων περιοχών και να το διαχειριστούν σωστά και δυστυχώς πιστεύω πως δεν μπορούμε καν να πούμε πως ένα κράτος μέλος έστω έχει ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια, που είναι πολύ λυπηρό, γιατί αυτή η νομοθεσία ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και έπρεπε να έχουν ε, υλοποιηθεί εδώ και πάνω από πέντε χρόνια. Ειδικά λόγω της κακής ποιότητας του αέρα σε αρκετές μεγάλες πόλεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 15 χρόνια μετά από την ε, ε, ημερομηνία επίτευξης των σχετικών στόχων. Επίσης, όσον αφορά την επεξεργασία αστικών λιμάτων, τα δύο τρίτα των κρατών μελών αντιμετωπίζουν ακόμα προκλήσεις με αυτή την, την, υπόθεση. Οι περισσότερες επενδύσεις χρειάζονται και η έκθεση δείχνει επίσης ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχουν για να βοηθήσουν για τις προσπάθειες εφαρμογής. Αυτό με φέρνει στο δεύτερο λόγο για τον οποίο αυτές, αυτή η έκθεση ε, ε, ε, εφαρμογής των περιβαλλοντικών νομοθεσιών έχει συνταχθεί. Πρώτον, για να δούμε πολιτικά που βρισκόμαστε. Δεύτερον, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε τη βοήθεια και την αρρωγή που μπορεί να προσφέρει η ε, Κομισιόν ε, με κονδύλια αλλά και με εμπειρογνωμοσύνη. Και έπειτα όταν εργαζόμαστε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ε, Εξαμήνου και την προετοιμασία του κράτους, των κρατών μελών του προγραμματισμού για τη χρήση των διαρθωτικών ταμείων στα επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τρίτος λόγος για τον οποίο εμείς προετοιμάζουμε αυτήν την έκθεση περιβαλλοντικής ε, εκτέλεσης εφαρμογής, αυτό ε, συμβαίνει ώστε να δώσουμε το ok στα κρατημέλη, ε, να τους πούμε ναι, ορίστε, έχετε να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση, να πούμε σε κάθε υπουργό περιβάλλοντος που ορίζεται στα 27-28 κρατημέλη, να, αυτό είναι εδώ το χαρτοφυλάκιό σου, έχεις μεγάλη πρόκληση, θα έρθει η Κομισιόν σε ένα, δύο, τρία χρόνια με διαδικασία κατά παράβαση. Μη με έρθει και μας πεις γιατί μετά από δύο χρόνια ή τρία χρόνια ότι ε, δεν το ήξερε. Εμείς σε προειδοποιούμε, υπάρχει αυτή η πρόκληση, πρόκληση και η πρόκληση είναι μεγάλη. Αφού όμως λοιπόν έχουμε δει και ελέγξει πώς και αν εφαρμόζονται όλα αυτά, θα ήθελα να είμαι σαφής. Μια συγκεκριμένη πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε οποιοδήποτε κράτος μέλος δεν μπορεί να εξαρτάται μόνο από την αστυνόμευση ή στην επιβολή κυρώσεων. Πρέπει επίσης να βασιστούμε στην πρόβλεψη, την προετοιμασία και την εργασία πριν να επιβληθούν πρόστιμα. Ε, και το κάνουμε αυτό με τα 28 κράτη-μέλη Έχουμε διμερή διάλογο με πολλά από αυτά, αλλά νομίζω πως θα ήταν εκτιμητέο ένα μήνυμα από εδώ, από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο στη διάρκεια αυτής της αιτίας, ένα ισχυρό μήνυμα για ε, ε, ενισχυμένο διάλογο ενώ μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών μελών για θέματα ε, εφαρμογής, γιατί δεν είναι μόνο ένα γραφειοκρατικό θέμα, ε, όταν ε, έρχεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου του Περιβάλλοντος, μετά από το νομιθετικό κομμάτι, οι υπουργοί φεύγουν και αρχίζουν να χρησιμοποιούν το κινητό τους και αντικαθίστανται από τους γενικούς τους γραμματείς, διευθυντές ή, εν πάση περιπτώσει, από τον μόνιμο εκπρόσωπό τους. Εάν πάρετε φωτογραφίες σε αυτή την αίθουσα, ε, αυτό συμβαίνει για πάνω από τα δύο τρίτα των κρατών μελών. Όμως η εφαρμογή, δηλαδή η απόδοση, η συγκεκριμένη που αναμένουν οι πολίτες και οι οικονομικοί φορείς είναι πολύ ε, σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή πρέπει να υιοθετούμε πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς ε, νόμους, αλλά το ίδιο σημαντικό είναι και το να αποδίδουν αυτοί. Αυτό περιμένουν οι πολίτες. Πραγματικά θα θέλαμε λοιπόν ένα μήνυμα τέτοιο ισχυρό. Και έτσι έρχομαι στο τέλος της παρουσίασής μου, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα το εκτιμούσαμε αν η Επιτροπή σα και το Ευρωκοινοβούλιο μπορούσαν να στείλουν μηνύματα για διάφορα οριζόντια ευρήματα τα οποία περιλαμβάνονται στο, στην οριζόντια ανακοίνωση που συνέταξε η Κομισιόν. Και το πιο σημαντικό σημείο, Πρόεδρε μου, ε, και επιτρέψατε μου να το τονίσω αυτό είναι ότι ακόμα και αν εφαρμόσουμε, μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε 100% με την νομοθεσία περί υδάτων ή με τη νομοθεσία περί φύσης ή περί ε, αέρα εάν οι δημόσιες πολιτικές σε άλλους τομείς ε, για το περιβάλλον δεν συντηριάζονται με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, εάν η γεωργική πολιτική, η ενεργειακή πολιτική, η πολιτική μεταφορών και η βιομηχανική πολιτική δεν είναι ευθυγραμμισμένε με την περιβαλλοντική πολιτική, δεν θα συμμορφωθούμε 100%. Αυτό δεν σημαίνει πω η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να έχει το πάνω χέρι σε σχέση με τι άλλε πολιτικέ. Όχι, αλλά θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε όλε αυτέ τις πολιτικέ, Γιατί αυτή τη στιγμή η γεωργική πολιτική, η πολιτική μεταφορών, η πολιτική για τα αστικά κέντρα που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι δεν είναι, μόνο δεν είναι βιώσιμε, αλλά ορισμένε είναι και δεν επιτρέπουν καλά ευρωπαϊκά ε, ε, περιβαλλοντικά με αποτελέσματα σε κάποιες περιπτώσεις. Να σας πω ότι και η ποιότητα της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γνωρίζουμε ένα από τα βασικά εμπόδια ανάμεσα στους ισχύοντες κανόνες, δηλαδή στα βιβλία, και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες και γιατί υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο τι λένε οι κανόνες και το ποια είναι η κατάσταση επιτόπου. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή τα προβλήματα είναι τεχνικά περίπλοκα μόνο, Ορισμένα ναι, είναι τεχνικά περίπλοκα, άλλα χρειάζονται περισσότερα χρήματα, αλλά και πολλά από αυτά απαιτούν πολιτική βούληση και ιδιαίτερα τη βούληση κανείς να εξασφαλίσει ότι σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ότι γίνεται συμμόρφωση με το νόμο. Και αυτό εξασφαλείται από τους εθνικές επιθεωρητές, από τους επιθεωρητές του υγειονομικού και ούτω καθεξής. Η διακυβέρνηση λοιπόν της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι εξίσου σημαντική. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ελπίζω να μην σας κούρασα και ε, βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια, προτάσεις ή ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Μιλήσατε με την καρδιά σας και με πάθος, όχι μόνο από γραφειοκρατική θέση. Το εκτιμάμε ιδιαίτερα. Ξεκινάμε το ΚΑΤΣΔΙΑΕ με τα μέλη με το έλκα ο κύριος Λουένα. Ε, ε, σοσιαλιστές κύριε Πρόεδρε, σοσιαλδημοκράτες, μικρή διαφορά. Λεπτομέρεια, μικρή λεπτομέρεια, αμεληταία. Λοιπόν, ε, για το, την ποιότητα του αέρα ε, είπατε 400.000 θάνατοι το ετησίω λόγω χρόνιων ε, ασθενειών που οφείλονται στη ρήπανση. Αυτό τα λέει το Ευρωβαρόμετρο. Μέσα στη διαδικασία αξιολόγηση της οδηγίας περιποιότητας του αέρα να μελετήσετε τη δυνατότητα ενό κανονισμού που υποχρεώνει τη δημιουργία ε, ζωνών άνευ κυκλοφορία οχημάτων, ας πούμε για την κεντρική Μαδρίτη ε, καταφέραμε να σταματήσουμε ε, την τρέλα αυτή που ήθελε να επιβάλλει η το, Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα θα συνεχιστεί αυτό το σχέδιο για το Μαδρίτη Σεντράλ, δηλαδή πεζόδρομο στην κέντρο της Μαδρίτης. Ε, η ιδέα του να τονιστεί το πρόβλημα του πολύ ε, μολυσμένου αέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συμφωνήσουμε όλοι και να δεσμευτούμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ από τους σοσιαλιστές λοιπόν. Και πάλι η κυρία Μαρία Αρενά. Ευχαριστώ. Έχω να μιλήσω σε, για τρεις τομείς. Ε, την εφαρμογή των εργαλείων της κυκλικής οικονομίας, πρώτον και τη διαχείριση των αποβλήτων. Τα εργαλεία που ψηφίστηκαν και πρέπει να εφαρμόσουμε στην Αλία, ε, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξάγει απόβλητα στο εξωτερικό. Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι σε αναπτυσσόμενες χώρες, ε, αφρικανικές όπως την Γκάνα ειδικότερα, βρίσκουμε ε, σκουπίδια ευρωπαϊκά στα, για παράδειγμα, ηλεκτρικές συσκευές. Έχουν λάβει τη μορφή μάλιστα δωρεών. Πρόκειται για παραβίαση, ε, για παράκαμψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να εφαρμόσουμε εργαλεία νομοθετικά ώστε να μην φτάνουν αυτές οι δωρεές ε, στις χωματερές στην Αφρική και στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε και για έγκλημα, μιλάμε για εγκληματικέ ομάδε που διοχετεύουν αυτά τα απορρίμματα σε αυτέ τι χώρε. Τι γίνεται λοιπόν από τα κράτη-μέλη και τα τελωνία ώστε να παρεμποδίσουμε αυτού του είδου παράκαμψη τη νομοθεσία. Το δεύτερο θέμα αφορά την νομοθεσία σε θέματα χημικών προϊόντων. Τι γίνεται σήμερα ούτω ώστε η νομοθεσία κατά των λοιπασμάτων ή των ενδικρινικών διατρακτών να μην φτάνουν μέσω της εξωτερικής παραγωγής. Έχουμε μιλήσει πολύ για το διεθνές εμπόριο στο πλαίσιο αυτού, αυτό που απαγορεύεται στην Ευρώπη μπαίνει από το παράθυρο. Μέσω των εμπορικών συμφωνίων πώς μπορούμε να το αποφύγουμε. Και το τελευταίο που ήθελα να πω αφορά την αποτελεσματικότητα. Είπατε προηγουμένω ότι είναι σημαντικό στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να συμπεριλάβουμε το περιβαλλοντικό ζήτημα. Πώς λαμβάνεται υπόψη αυτό στα μεταρρυθμιστικά σχέδια. Πώς ε, μια περιβαλλοντική επένδυση μπορεί να μην εντάσσεται στον κανόνα του 3% και του 15% της ε, δημοσιονομικής ε, ε, στάθμισης. Πρέπει να γίνει αυτό. Πρόκειται για επενδύσεις. Σας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα εργαλεία ευελιξίας στον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε βιώσιμες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Κάτι που βγαίνει εκτός αρμοδιότητων του αρμοδίου που έχουμε εδώ μπροστά μας. Για το ΕΛΚΑ ε, εξακολουθεί να μην υπάρχει κάποιο ε, Για το ΡΙΝΙΟΥ η κυρία Πόβη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και του συναδέλφου από την Κομισιόν. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, λέει η κυρία Μπρόφη. Αυτή η αναθεώρηση είναι μια καλή διαδικασία. Την υποστηρίζουμε ώστε να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να επιταχύνουμε την υλοποίηση, χωρί την οποία δεν έχει νόημα να έχουμε φιλόδοξους ε, περιβαλλοντικού κανόνες αν τα κράτη-μέλη δεν κάνουν τη δουλειά τους, οι πολίτες τους είναι οι ίδιοι αυτοί που υποφέρουν. Οι συστάσεις της Κομισιόν μας βοηθούν πολύ, αυξάνουν τη διαφάνεια, επισημαίνουν και τις βέλτιστες πρακτικές από τις οποίες μπορούν να μάθουν όλα τα κράτη-μέλη. Ενθαρρύνουμε λοιπόν την Κομισιόν να συνεχίσει τη διαδικασία. Ταυτόχρονα όμως η έκθεση δείχνει ε, κάτι ανησυχητικό τεράστιες διαφορέ ε, στον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνουν τα καθήκοντά του τα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη-μέλη απλά δεν ασχολούνται. Δεν εφαρμόζουν τίποτα. Είναι σημαντικό λοιπόν νομικά να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ω θεματοφύλακα ε, τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, Να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ξεκινώντα διαδικασίε επί παραβάση ε, έναντι κρατών που παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πώς βλέπετε τη σχέση μεταξύ τη αναθεώρησης και ε, των πόρων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι δεν αποδυναμώνει τη στάση της για τις διαδικασίε επιπαραβάσεις η Κομισιόν, αλλά ότι θα δείξει μεγαλύτερη αυστηρότητα, λαμβάνοντας δράση κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία. Και τέλος, όσον αφορά συγκεκριμένα προβλήματα, η ποιότητα του αέρα στη δική μου τη χώρα, των ΗΠΑ Βασίλειο, είναι σοβαρό πρόβλημα. Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε πληροφορίε από την εμπειρία σα, πώ μπορούν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και τι κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, πράσινη, παρακαλώ. Η κυρία Πάολο, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για αυτέ τι σημαντικέ πληροφορίε που μα έδωσε η Κομισιόν. Η αναθεώρηση αυτή είναι πολύ σημαντική. Απογοητεύομαι που αντιλαμβάνουμε ότι η βιοπικιλότητα και το περιβάλλον υποφέρουν ακόμη περισσότερο παρότι έχουμε φιλόδοξη νομοθεσία. συνέκρινα λίγο με την έκθεση του 2017 και μεταξύ των, της έκθεσης 2017 και 2019. Και θεωρώ ότι το θέμα είναι, το ερώτημα είναι πώς βοήθησε η έκθεση να βελτιωθεί η υλοποίηση, γιατί τα προβλήματα είναι τα ίδια. Κατά την άποψή μου, ο κατάλογος των κρατών μελών που δεν έχουν ε, προβεί σε επαρκή υλοποίηση μεγαλώνει και το χάσμα διευρύνεται. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την αναθεώρηση, την έκθεση, τη δράση, ούτω ώστε να γίνει πιο βιώσιμη η κατάσταση και να έχει περισσότερο νόημα. Και το άλλο που τονίσατε ότι το σημαντικότερο είναι ότι η περιβαλλοντική πολιτική δεν έχει ενταχθεί σε άλλες πολιτικές, δεν έχει ενσωματωθεί και συνήθως πρέπει να κάνει πίσω. Ε, Προ όφελο οικονομικών ζητημάτων, οδικών ζητημάτων, υποδομών, οδικών υποδομών κτλ. Κατά την απόψή σα τα κράτη-μέλη κατανοούν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Έχουν θεσπίσει δομές όπως ε, συζητήσεις ε, των Υπουργών σε περιβαλλοντικά θέματα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει, να γίνονται κατά την άποψή μου τους, ώστε να μην μένει πάντα ε, στην τελευταία θέση το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το ID κυρία Μπενιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα καθημερινό, καθημερινό πρόβλημα με απασχολεί το καλοκαίρι. Είχαμε ελλείψεις φαρμάκων στη Γαλλία. Η μετατόπιση των παραγωγών καθυστερεί τη δρομολόγηση των προϊόντων. Επίσης, εργαστήρια στην Κίνα ε, παράγουν ε, περισσότερο για τη Γαλλία διότι θεωρούνται πιο αποδοτικά οικονομικά. Είναι σκάνδαλο. Τον Ιούνιο 2.318 φάρμακα έλειπαν, ε, παρουσίασαν ελλείψει και αργότερα πλασιάστηκε αυτό. Ένα στου τέσσερι Γάλλου αντιμετώπισε το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό θέμα. Αυτή η έλλειψη είναι ενισχυτική. Το 80% των δραστικών ουσιών παράγονται εκτό Ευρώπη σε σχέση με το 20% πριν από 20 χρόνια. Ένα ε, ασθενή, για παράδειγμα, που υποφέρει από καρκίνο δεν μπορεί να καθυστερεί τη θεραπεία του, διότι ορισμένε φαρμακοβιομηχανίε ασχολούνται με την ε, κερδοφορία του. Οι ε, θεραπείε πρέπει να είναι προσβάσιμε σε όλου. Προτείνω, κύριε Πρόεδρε, να ε, εξετάσετε αυτή τη μετατόπιση της παραγωγής των ε, φαρμάκων, να δείτε πώς θα την αντιμετωπίσετε με φοροαπαλλαγές ενδεχομένως στη φαρμακοβιομηχανία ή με κάποια εξέλιξη των στρατηγικών αποθεμάτων. Ευχαριστώ. The last question ε, from the... Ευχαριστώ. Η τελευταία ερώτηση, σοσιαλδημοκράτες, κυρία Γκιούτελαντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Κομισιόν που βρέθηκε σήμερα εδώ μαζί μας και που είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα μαζί της που αφορά τους πολίτες και, τους, ε, και τις ζωές τους. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την ποιότητα του αέρα. Συμφωνώ με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Λουένα, για την ε, σημασία αυτού του σοβαρότατου προβλήματος που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της να καταστήσει το θέμα αυτό μεγαλύτερη προτεραιότητα και να συνδέσει όλους τους ε, τομείς πολιτικής που αφορούν στο περιβάλλον και να κατατείνουν όλες τις προσπάθειες στην ε, βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις. Για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται καλή συνεργασία με τους μεγάλους παίκτες που βρίσκονται στις μεγάλες, ε, στις μεγάλες ιδίως πόλεις, στα μεγάλα αστικά κέντρα γιατί νομίζω ότι μια τέτοια διαδικασία θα είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι Δήμοι, όλες οι μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη θα θέσουν το θέμα της ποιότητας του αέρα ως ύψιστη προτεραιότητά τους, ακριβώς λόγω του ότι αυτό θα προκύπτει και από τα πάνω, από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τα θέματα που έθεσαν. Επειδή ε, τέθηκαν και ορισμένα ζητήματα αρχής. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πολύ σοβαρή την εφαρμογή των ε, ισχυών των κανόνων. Πράγματι, υπάρχουν κενά στην ε, υλοποίηση, στην εφαρμογή και καταβάλουμε κάθε ε, δυνατότητα που έχουμε, κάθε αρμοδιότητα επιβολής των κανόνων και υπάρχει ξεχωριστό στο, ε, μάλιστα στο, στην υπηρεσία περιβάλλοντος της Κομισιόν ε, από την υπηρεσία αυτή έχουν ξεκινήσει οι περισσότερες διαδικασίες επί Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να βασίζεται μόνο στην επιβολή των κανόνων γιατί όταν υπάρχουν τόσο πολλές παραβάσεις ε, είναι λογικό να συμπεράνει κανείς ότι υπάρχουν και κάποιες παθολογίες, κάποια, κάποια στοιχεία, κάποια προβλήματα εν γενή αν θέλετε και αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και απαντώ και με αυτό στον συνάδελφο από τους Πρασίνους. Τι κάνετε για την καλύτερη εφαρμογή ήταν το ερώτημά του. Εμείς στην αναθεώρηση της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής έχουμε δημιουργήσει ένα εργαλείο peer-to-peer μεταξύ ομοτήμων. Δηλαδή, στέλνουμε εμπειρογνώμονες από τη μία χώρα σε άλλη χώρα. Για να μην χρειάζεται να ξαναανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή. Όταν και όπου έχει προσδιοριστεί σε κάποιο κράτο μέλο μια πολύ ευφυή λύση, για παράδειγμα, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, των λιμάτων, για την βελτίωση τη ποιότητα του αέρα, αυτέ οι λύσει μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλα κράτη-μέλη. Και ε, τα κράτη-μέλη έχουν πραγματικά εκφράσει την ε, πολύ βαθιά εκτίμησή τους για τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε. Είναι εξαιρετικές οι λύσεις που μπορούν έτσι να αξιοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πάνω από 50 σχετικές εκδηλώσεις έχουμε ε, διοργανώσει. Χωρίς καθόλου να πειράξουμε την νομοθεσία. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα διαρθρωτικά ταμεία για να συνδράμουμε είτε την ε, καινοτομία και τις ε, καινοτόμες λύσεις, είτε τις επενδύσεις σε σκληρές υποδομές. Πρέπει όμως να σας πω ότι βαθμιαία τα τελευταία 10 χρόνια τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν εξελιχθεί με τέτοιον τρόπο ώστε όλο και λιγότερα λεφτά διατίθενται προς τις σκληρές ε, υποδομές, τις παραδοσιακές δηλαδή, και όλο και περισσότερα χρήματα κατευθύνονται στις στις καινοτόμες λύσεις. Να το έχετε και αυτό υπόψη σα. Και το ξέρουν και τα κράτη-μέλη. Πολλοί ευρωβουλευτέ έθεσαν το ζήτημα της ε, μόλυνσης του αέρα. Ιδίω σε αυτό το τομέα έχουμε συνεργαστεί στενά με ε, τα κράτη-μέλη, έχουμε δει πολλέ ενδιαφέρουσες ευφυεί λύσει σε πολλούς δήμους. Είδαμε όμως και πολλές λύσεις που έχουν μόλις πρόσφατα ε, εφαρμοστεί και προφανώς δεν έχουν ακόμα αποφέρει τα αποτελέσματα. Έχουμε προσφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον κρατών ε, μελών και πολλά έχουν καταδικαστεί για λόγους ρήπανσης του αέρα. Όμως αυτός δεν είναι ο τελικός μας στόχος. Στόχος μας δεν είναι να καταδικάζονται τα κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα του αέρα και γι' αυτό το σκοπό συνεργαζόμαστε με, πολλά, με τα κράτη-μέλη και πολλοί δήμαρχοι έχουν πράγματι ε, βρει πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις. Επίσης, ε, βρισκόμαστε σε έναν διάλογο για τον καθαρό αέρα με τα κράτη-μέλη και προσπαθούμε να εμπλέξουμε και τις τοπικές αρχές οι οποίες είναι αναντικατάστατες γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να θεσπίζουμε κανόνες από τα πάνω το θέμα είναι πώς ακριβώς θα εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες και στον τομέα της, ε, του, της ρήπανσης του αέρα οι δήμαρχοι είναι αυτοί που πραγματικά καλούνται να εφαρμόσουν πρακτικά μέτρα. Κυρία Αρενά, θέσατε μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα θα, βάλω, θα σας απαντήσω μαζί για την κυκλική οικονομία και τα χημικά προϊόντα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που ε, είπατε. Και πράγματι δεν μας περιποιεί η τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση αυτή. Έχουμε κανόνες στον ΟΑΣΑ και αυτοί οι κανόνες έχουν υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαγορεύεται στα κράτη-μέλη να εξάγουν μη ε, διαχωρισμένα ε, απορρίμματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο γίνεται πολύ συχνά. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται απορρίμματα ε, από την Ευρω... που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που δεν έχουν υποστεί κάποια ε, διαδικασία διαχωρισμού. Αυτό άλλωστε ήταν και ο λόγο για τον οποίο η Κίνα απαγόρευσε τι αγωγέ απορριμμάτων. Έχουμε βρει σε άλλε περιπτώσει αντίστοιχα φορτία απορριμμάτων από την Ευρώπη και στην, ε, από, ε, Αφρική. Εδώ ε, ο, λόγο, ο τρόπος για την αντιμετώπιση ε, βεβαίως είναι η ενίσχυση των ελέγχων. Οι τελωνιακέ αρχέ πρέπει να ενισχυθούν. Φανταστείτε ότι μόλις το 5% των εισαγωγών χημικών προϊόντων ε, έχει καταστεί δυνατό να ε, ελεγχθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αθέμητο ανταγωνισμό που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό REACH από παραγωγούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα από τα βασικά θέματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και που θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο των μελλοντικών μας πολιτικών ενάντια στα φυτοφάρμακα, τη χημική ε, μόλυνση και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες θα είναι η βελτίωση του ελέγχου της αγοράς προκειμένου να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, επειδή κάποιος ε, ρώτησε και στον τομέα αυτό τη σχέση μας με τους δημάρχους, ε, σκεφτόμαστε να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτή την πλατφόρμα, ε, την Σύνοδο των Δημάρχων, για να μπορέσουμε και εκεί να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Και τελικό ερώτημα, τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν και τι δεν μπορεί να κάνει η Κομισιόν. Εμείς μπορούμε μέσω των διαδικασιών παραβάσει να κάνουμε πολλά. Έχουμε το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο και αυτό λέει πολλά, γιατί ε, προηγήθηκε πολύ μεγάλο ε, έργο. Ωστόσο δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα φυσικά. Σας το λέω ειλικρινώς και έτσι οφείλω να σας μιλώ ειλικρινώς. Φυσικά, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι άπειρα. Υπάρχει όμως ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας που υπάρχει. Η πρόσβαση στην δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη-μέλη και μία από τις προτεραιότητες της Κομισιόν τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι να εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τη λειτουργία αλλά και την πρόσβαση ε, στα εθνικά δικαστήρια που χειρίζονται περιβαλλοντικές υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε στο τέλος της συνεδρίασής μας τώρα και θα τα ξαναπούμε στις 25 Σεπτεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Θα τα ξαναπούμε εκείνη την ημερομηνία. Ευχαριστώ.